Περνάμε στις ψηφοφορίες σημείο 7 της ημερήσιας διαταξη αφού έχει ακυρωθεί η ψηφοφορία για τα δύο προηγούμενα. Πρόκειται για την ψηφοφορία τη ενδιάμεση έκθεσης του Ράιμερ Μπέγκε για το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2010 Ο Πρόεδρος Διακόπτη, παρακαλώ να σταματήσετε τι μεταξύ σα συζητήσει. Όλοι έχετε του καταλόγους ψηφοφορία ρωτήσω από τους εισηγητές αν θέλουν να πούν δύο λόγια. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Πρόεδρα πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε το στρατηγικό στόχο με αυτή την ενδιάμεση έκθεση. Τον έχουμε ήδη συζητήσει αυτόν και έχουμε συμφωνήσει εν ώψη της ε, προσαρμογής ε, του ε, πολιτού σε χρηματιστικού πλαισίου και της συμφωνίας, ε, κυρίως μετά τη θέση ισχύ της ε, συνθήκης Λισαβόνας, βρισκόμαστε σε μια μετέωρη κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό με αυτή την ενδιάμεση έκθεση να εμφανιστούμε στην Ολομέλεια, έτσι ώστε να εκπέμψουμε ένα ευκρινές μήνυμα απέναντι στην Κομισιόν και το Συμβούλιο. Θα ήθελα λοιπόν να πω για άλλη μια φορά ότι βλέποντας τις ε, τροπολογίες θέλω να σας προτείνω το εξής. Είμαι πρόθυμος να δεχθώ όλες τις ε, τροπολογίες υπό την προϋπόθεση ότι οι σημαντικές προτάσεις α και β θα ενταχθούν στο πακέτο. Δηλαδή παρετούμε από τις 2 ε, και 4 σε ξεχωριστή ψηφοφορία και στην τροπολογία 8 ε, προτείνω ε, να γίνει αποδεκτή. Και κάτι άλλο, αν τελικά περάσει αυτή η έκθεση, είναι σαφές ότι την Τρίτη στην Ολομέλεια θα γίνει η τελική ψηφοφορία. Και η τάση που επιδιώκουμε κατ' ουσίαν είναι έκκληση προς την Κομισιόν να αναβαθμίσει πολιτικά τις τεχνικές προδιαγραφές με την έννοια της μεγαλύτερης ευελιξίας, της διατήρησης, της αναθεώρησης, δυνατότητα αναθεώρησης που έχουμε σήμερα και ως εκ τούτου μέχρι το 2013 το όλο θέμα να έχει ε, μπει πάνω σε μια καινούργια βάση. Και ε, επιμένω κύριε Πρόεδρε στο ίτερ θα επανέλθουμε και θα πούμε επιτέλους η Κομισιόν να κάνει μια σοβαρή ανάλυση το τι ακριβώς ε, θα συνεπάγονται τα διάφορα προγράμματα μέχρι το 2013 σε επίπεδο χρηματοδότησης. Τι, τι κονδύλια θα χρειαστούν. Ε, και μόνο έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε μία μακροπρόθεσμα υπεύθυνη πολιτική. Νομίζω λοιπόν ότι για να το προβάλλουμε αυτό χρειαζόμαστε την ενδιάμεση έκθεση. Μάλιστα. Υπάρχει μια σειρά από τροπολογίε. Ο εισηγητή είναι σύμφωνο με όλε τι τροπολογίε. Μήπω αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να τι ψηφίσουμε αν μπλοκ ή όχι. Υπάρχουν αντιρρήσει. Το έλεγε συμφωνεί. Όχι, όχι. Οι φιλελεύθεροι διαφωνούν, οπότε δεν τα ψηφίζουμε αν μπλοκ Μάστε. Ναι, Άννα. Θέλουμε ψηφοφορία για την τροπολογία 4, χωριστή. Η Άννα ζητά να ψηφίσουμε χώρια την 4 μόνο. Για όλες τις άλλες μπορούμε unblock. Μάλιστα. Λοιπόν, ψηφίζουμε όλες τις τροπολογίες εκτός από την 4. Όλες οι τροπολογίες εκτός από 4 συμπεριλαμβανομένων και των συμβιβαστικών του εισηγητή, εκτός από την 4. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δύο κατά. Αποχές. Δεν υπάρχουν αποχές. Ωραία. Για την 4. Θέλετε χωριστή ψηφοφορία. Όχι. 4. Unblock. Ποιοι είναι υπέρ. Σας ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Τρεις αποχές. Εγκρίνατε λοιπόν. Σας ευχαριστώ. Η έκθεση του Ράιμερ εγκρίνεται λοιπόν. Α, ναι, πρέπει να κάνουμε και τελική ψηφοφορία. Λοιπόν, τελική ψηφοφορία. Όπως τροποποιήθηκε η έκθεση, είναι υπέρ. Κατά. Δύο. Αποχές. Δύο κατά. Καμία αποχή. Ωραία. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Και έτσι αυτό θα γίνει αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης της δεύτερης ολομέλειας Σεπτεμβρίου, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα. Επόμενη ψηφοφορία. Έκθεση του κυρίου Καλφίν. Σημείο 20. Pardon. Euh, c'est, pardon. Il y a d'abord le budget Όχι, συγγνώμη. Διορθωτικός προπολογισμό. 5. Πού είναι? Ο προϋπολογισμός που αφορά την ΟΛΑΦ. και την προσαρμογή των πόρων ε, που σχετίζονται με το προπολογισμό ΟΛΑΦ. Ήδη είχαμε ακούσει η παρουσίαση του εισηγητή, όπως μας το είχε πει ο Λάζλος Σουριάν και βέβαια μπορούμε να διορθώσει αν κάνω λάθος. Όπως κάναμε πολλές φορές, πρόκειται για μια ψηφοφορία προληπτική που δεν θα διαβιβάσουμε στα υπόλοιπα θεσμικά όργανα παρά μόνο όταν το Συμβούλιο θα έχει από τη μεριά του εκφραστεί. Λάσλο Σούρια, αν θες να πεις κάτι ή να ψηφίσουμε αμέσω. Δεν έχεις να πεις τίποτα. Ωραία. Υπέρ. Υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Ένας κατά. Αποχές. Καμία αποχή. Εγκρίνεται. Το ίδιο και για το 19. Σχέδιο δοστικού προϋπολογισμού επαριθμών 7. Το έχουμε συζητήσει επί μακρόν, δις. Κανονικά το Συμβούλιο θα πρέπει να υιοθετήσει τη θέση του στη διάρκεια της ημέρας και άρα και εδώ είναι μια προληπτική ε, ψηφοφορία. Ο κύριος Συγητής έχει το λόγο. Είμαι πάρα πολύ σύντομος πρόεδρε. Υπάρχει τεχνικό πρόβλημα, δεν ακούγεται ο μίλητης. I that νομίζω ότι η πραγματική επιτυχία της Επιτροπής μας και του Κοινοβουλίου γενικότερα και συγκεκριμένα ημών, πρόεδρε, που προτείνεται αυτή την ε, πρόταση και αυτή την επιθυμία να περιληφθεί αυτό το κονδύλιο του ώστε να επιληθεί το πρόβλημα αλλά και να καταστεί εφικτόν το κοινοβούλιο να συμμετάσχει σε όλο αυτό το σχέδιο διάσωσης. Και λοιπόν πάρα πολύ ότι μόλις σήμερα κυκλοφόρησε το τελικό κείμενο όμως επανειλημμένα το συζητήσαμε στην Επιτροπή μας. Αλλά και στον ε, τριμερή διάλογο, στον τριμερικό διάλογο, να μην έχουμε άλλες ε, παρελκύσεις και έτσι να μπορέσουμε να αποκρισταλώσουμε κάποια θέση. Άρα παρακαλώ συνάδελφοι να στηρίξετε αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ κύριε Ζήκητα Και τώρα θα ψηφίσουμε τον διορθωτικό προηγούμενο των 7. Ποιοι είναι υπέρ. Σας ευχαριστώ. Ποιοι είναι κατά. Δύο. Δεν έχουμε ε, αποχές και επομένως εγκρίνεται ακριβώς από τους όρους που είπαμε και προηγουμένως. Και τώρα μπορούμε να πάμε στο σημείο υπαριθμών 20, δηλαδή την τροποποίηση του κανονισμού 1905 που αφορά την θέσπιση ενό μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας. Πρόκειται για την έκθεση Κάλφιν. Έχετε τον κατάλογο της ψηφοφορίας. Έχουμε πέντε τροπολογίες. Μήπως θέλει κάτι να πει ο συγκητής. Δεν είστε υποχρεωμένος. Όχι, σιωπά. Επομένω. μπορείτε λοιπόν, να τις ψηφίσουμε όλε μαζί. Ποιοι είναι υπέρ Ευχαριστώ. Ποιοι είναι κατά. δύο Αποχές. Δεν έχουμε αποχές. Επομένως εγκρίνεται. Και σας ευχαριστώ. Πρέπει να γίνει και άλλη μια συνολική ψηφοφορία. Μάλιστα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Μπάρμπαρα, είστε υπέρ ή κατά favorable, υπέρ, ωραία. Η διόπτωση ψηφοφορία, πάρα πολύ λογικό, συνεπές και τώρα μπορούμε να πάμε εις το θέμα που αφορά τις μεταφορές πιστώσεων. Σούριαν και Ρόμπιν Μάνκα. Oui. Can you specify which uh, is to be voted. transfer? Ε, νομίζω ότι για το 40 πρέπει να ψηφίσουμε. 40 κάτω 2010. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ πήγον θέμα. Το Πακιστάν πρέπει να βοηθήσουμε. Μάλιστα σωστά. Αυτό είναι η συνέχεια για την βοήθεια προς το Πακιστάν. Α, όχι, λέει διορθώνει πρόεδρος. Το 40 είναι το Σουδάν. Ε, ε, ε, ναι, δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Όχι, το Πακιστάν δεν είναι το Σουδάν, αλλά το πρόβλημα είναι ότι είναι επίγον θέμα και το υποστηρίζω. Οι δύο αυτές χώρες υποφέρουν από διαφορετικές τραγωδίες, αλλά που συμβαίνουν ταυτόχρονα. Και τα δύο έγιναν το καλοκαίρι. Πολύ επίγον. Σουδάν είναι η μεταφορά 40 και το Πακιστάν που είναι το 49. Αυτά. Λοιπόν, ψηφίζουμε λοιπόν για την 40. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δύο εποχές. Δύο εποχές λοιπόν ε, εγκρίνεται. Τώρα, 36. Μπορούμε να το εγκρίνουμε σήμερα, αν είναι έτοιμο. Άλλιως το ψηφίζουμε άλλη φορά. 36 για την Όλαφ. OK. Donc on le soumet au vote. Qui est pour l'amendement, le, le virement 36 Είναι υπέρ της μεταφοράς 36. Ευχαριστώ, κατά. Ευχαριστώ. Αποχές. Α, εγκρίνεται. Όσον αφορά τα άλλα θεσμικά όργανα, χρειάζεται να ψηφίσουμε επίσης το ΣΕ8 του Κοινοβουλίου. Ο εισηγητής μας, ο κύριος Μάνκα, είναι εδώ. Μάλιστα βρίσκεται μπροστά μου. Κύριε εισηγητά. Θα ήθελα να πω ότι πρόκειται για μεταφορά κονδυλίων στο C8. Πρόκειται λοιπόν για μια, ένα αίτημα να αυξηθεί αυτό το κονδύλι για τις ε, λειτουργικές ε, δαπάνες ε, του Γραφείου Ταξιδίων. Ε, υπήρξε κάποια διαδικασία επιλογής, αλλά δεν εντάχθηκε το ποσό αυτό στον προπολογισμό και εγώ προτείνω τώρα να το δεχτούμε. Ευχαριστώ. Πληρω... Ε, ψηφίζουμε, συγγνώμη, το σε 8 λοιπόν, τη μεταφορά σε 8. Υπέρ, κατά. Ευχαριστώ. Αποχές. Εγκρίνεται. Στη συνέχεια έχουμε τέσσερις τροπολογίες ε, του ελεγκτικού συνεδρίου, κύριε Σιγητά. Έχουμε λοιπόν ε, τέσσερις μεταφορές κονδυλίων ε, σε σχέση με το ελεγκτικό συνέδριο. Ε, το ένα είναι η οριζόντια, το οριζόντιο αποθεματικό 5%, ένα απόθεμα σε κάθε οργανισμό που έχει μεταφραστές. Το συζήτησαμε ήδη την τελευταία φορά. Εγώ προτείνω να αποδεσμευτεί αυτό το αποθεματικό του 5%. Ωραία, είναι η τροπολογία 1. Ναι, το 1. Ίσως να μας το παρουσιάσετε και τα 4 για να, τις 4 για να ψηφίσουμε μπλοκ. Πολύ ωραία λοιπόν. Πάμε στην 2. Το Μάιο έξι μέλη του ελεγκτικού συνεδρίου, εγκατέλειψαν την υπηρεσία και προσθέθηκαν έξι καινούργια μέλη. Αυτό συνεπάγεται κάποιες δαπάνες. Αυτό ήταν το δύο. Τώρα, στο τρία πρόκειται για την ενίσχυση κονδυλίων σε σχέση με τη συντήρηση των κτηρίων. Δεν πρόκειται για μεγάλο ποσό, προτείνω να το δεχτούμε. υπάρχουν τέσσερα... Εδώ δεν πρόκειται για μεγάλο κονδύλι, πρόκειται για ποτά αναπτυκτικά κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων, για έπιπλα και πρόκειται και για εξοικονόμηση σε σχέση με άλλα κονδύλια. Μας εγώ προτείνω να δεχθούμε και τα τέσσερα αυτά σημεία. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ. Η συγκεκριτής είναι υπέρ αυτών των τεσσάρων μεταφορών που μας εξήγησε την αιτιολόγησή τους και άρα σας προτείνω να τα ψηφίσουμε unblock. Ποιοι είναι υπέρ αυτών των τεσσάρων μεταφορών. Ευχαριστώ. Κατά. Δύο αποχές. Καμία αποχή. Εγκρίνονται λοιπόν και οι τροπολογίες του ελεγκτικού συνεδρίου. Και τώρα πάμε στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο. Εδώ υπάρχουν τρεις μεταφορές. Εδώ στο Κομπονιούς αναφέρονται δύο, αλλά ε, από ό,τι μου λένε υπάρχει και μία μεταφορά του άρθρου 47. Μπορείτε να μας τα παρουσιάσετε και τα τρία κύριε Σιγητά. Λοιπόν, εδώ έχουμε αυτές τις μεταφορές λόγω του ότι την τελευταία φορά τις απορρίψαμε. Ε, είχαμε άλλη μια συνεδρίαση πριν από τις διακοπές. Είχαμε μεταφορά κονδυλίων ε, σε σχέση με τις μεταφράσεις, ε, κυρίως αυτές της ΟΚΕ και της Επιτροπής των Περιφερειών. Σήμερα εγώ πήρα ένα ηλεκτρονικό μήνυμα, ίσως και εσείς συνάδελφοι, όπου αναφέρεται ότι ορισμένα πράγματα δεν αναφέρονται στο κόμπου νιούς. Ε, τεχνικό είναι το λάθος. Εμείς αυτό το θέμα το είχαμε συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξη του Ιουνίου και προτείνω οι μεταφορές αυτές ε, να γίνουν αποδεκτές. Μεταφορές ε, του Οικονομικού και Κοινωνικής Κοινωνικής Επιτροπής, ε, της Επιτροπής των Περιφερειών, Κοινοβουλίου, ε, Κομισιών και αυτά έχουν σε σχέση με το αποθεματικό του 5% για τις μεταφράσεις. Πολύ καλά λοιπόν και σας ευχαριστώ για αυτή την επιφύλαξη που είχατε ζητήσει. Επιτυχώς. Από το Συμβούλιο. Άρα τώρα θα ψηφίσουμε τρεις τροπολογίες. Ποιοι είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Άρα αυτά τα τρία κονδύλια για την ΟΚΕ έχουν εγκριθεί, επομένως δεν έχουμε τίποτε άλλο για τα θεσμικά όργανα και έχουμε ακόμη δύο ψηφοφορίες όσον αφορά το 23 της μερικής διατάξεως, δηλαδή την κτηριακή πολιτική. Συγκεκριμένα κυρία Χόλμαϊερ. Θα θυμάστε ότι υπήρχε ένα πρόβλημα όσον αφορά το έγγραφο στην Στοκχόλμη και επίσης υπήρχε πρόβλημα ε, της ε, ανακατασκευής του κτηρίου μας στην ΑΕΤ. Έχετε το λόγο συνάδελφα. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητέ πρόεδρε, πρώτα απ' όλα ε, θα ήθελα να ξεκινήσω με τη Στοκχόλμη στην Στοκχόλμη την παρουσίασα με λεπτομέρειε, ήδη κατά την τελευταία φορά, γι' αυτό δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Να σας αναφέρω μόνο ε, τα βασικά θέματα, ε, γιατί στην περίπτωση αυτή πρέπει να τοποθετηθούμε. Ο λόγος λοιπόν είναι ότι ε, τάξη, το κτίριο είναι θαυμάσιο και διαθέτει την ε, τελευταία τεχνολογία, ε, λειτουργεί με εξοικονόμηση ενέργειας, μόνο που κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας προέκυψαν κάποιες παρατυπίες, γιατί είχαμε δεχθεί μία συμφωνία όπου ε, πλέον δεν μπορούμε να αποφασίσουμε. Δηλαδή, αν έπρεπε να εγκαταλείψουμε το κτίριο, θα πληρώναμε τόσα πολλά πρόστιμα που κάτι τέτοιο θα ήταν σχεδόν αδύνατο. Και γι' αυτό λοιπόν ε, μια θολή σύμβαση η οποία προκύπτει χωρίς την δική μας ε, την έγκριση, γιατί τότε δεν ζητήθηκε η άποψη της Επιτροπής Προβλησμών. Αυτό είναι κάτι πολύ προβληματικό, γιατί με αυτόν τον τρόπο κατ' ουσίαν καταργεί κανείς το άρθρο 109. Το Κοινοβούλιο δεν μπορεί πλέον να αποφασίσει αν ισχύσουν όλα αυτά. Ε, και επίσης, ε, πάω τώρα στο επόμενο, φτάνουμε για το πρώτο. Για την IT θέλω να προσθέσω ότι Προφανώς εκεί δεν μπορούσαν να γίνουν διαγωνισμοί, ε, ούτε μεγάλη διαδικασίες. Μα ε, πού να γίνει διαγωνισμός, πώς να προκηρυχθεί και ποιο να συμπεριληφθεί. Ε, τα κτίρια είναι τόσο πολύ κατεστραμμένα που οι συνεργάτες μας εργάζονται στα σπίτια τους. Άρα δηλαδή για να υπάρξει λειτουργικότητα θα πρέπει να αναγερθούν νέα κτίρια. Νομίζω ότι η διαδικασία που εφαρμόζει εδώ η Κομισιόν είναι λογική, ρεαλιστική και εξυπηρετεί την αντιπροσωπεία στην IT. Κατά τα άλλα, ε, το κτίριο αυτό έχει 45 θέσεις εργασίας, ε, προβλέπονται δαπάνες ε, της τάξης των 3,7 εκατομμυρίων ευρώ και η αποζημίωση ή επαλωτρήσει 178.000. Αυτά τα ποσά θα διατεθούν σε δόσεις. Η επαλωτρίηση 178000 αυτα δόση θα είναι της τάξης των 18.700 ευρώ. Ε, δεν θέλω να μπω σε όλες τις γραμμές. Νομίζω τα πράγματα εδώ είναι ξεκάθαρα και συμφωνώ. Δέχομαι. Εισηγήτρια, ευχαριστώ. Όχι εκατομμύρια, δισεκατομμύρια. Είναι η τάξη μεγέθους. Ποιο είναι το σωστό. Oui, εκατομμύρια συνολικά. 18.700, <laughs> ε, μιλάμε εδώ για ε, τα προηγούμενα ψωά και όχι για εκατομμύρια. Λοιπόν, θα έγινε ένα λάθος ε, με του αριθμού. Κοιτάξτε, ίσως ε, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει μία απόφαση με ε, λογικές ε, αποφάσεις. Ε, συμφωνώ με αυτά που ελέγχθηκαν στο 1, 2, 3. Αυτά είναι πολύ καλύτερα. Πάντως δεν πιστεύω ότι πρέπει να υπερψηφίσουμε. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι ένα παράδειγμα όπου τα πράγματα πάρα πολύ γρήγορα μπορούν να πάνε και πολύ στραβά. Η συγκήτρια. Εγώ θα ήθελα απλά να επισημάνω ε, ότι εάν ε, δεν συμφωνήσει θα προκληθούν και πάλι δαπάνες και αν συμφωνήσει πάλι θα έχουμε δαπάνες μόνο ε, που δεν θα έχουμε καμία αποζημίωση. Γι' αυτό λοιπόν γκρά συντάξαμε αυτή τη γνώμη. Ευχαριστώ. Οπότε ψηφίζουμε. Πρώτα πρώτα. Άρθρο 179 όσον αφορά την έγκριση ε, για το κτίριο ε, του Κέντρου Πρόληψης Ελέγχου Νόσων. Είναι αυτό το οποίο ε, προτείνει η που Είναι υπέρ. Σηκώστε το χέρι. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ. Επομένως αποφασίζουμε να μην γνωμοδοτήσουμε. Όχι, όχι, όχι, όχι. Ναι, ναι, ναι, το, το ανάποδα λέει ο πρόεδρο. Το δεχθήκαμε, δεχθήκαμε. Και για την αντιπροσωπεία στην ΑΕΤ είπαμε ότι θα γνωμοδοτήσουμε και ε, είπαμε ότι γνωμοδοτούμε θετικά. Ε, γιατί πρώτη για το άρθρο 179 ε, είναι κατεπήγον και λέει η συγκήτρια να μην, να μην, να μην αποφανθούμε. Ποιο είναι υπέρ αυτού που είπε η συγκήτρια να μην αποφανθούμε για την ΑΕΤ. Σηκώστε το χέρι. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Μία αποχή. Άρα δεν θα ισχύσει το άρθρο 179 όσον αφορά το κτίριο για την αντιπροσωπεία στην IT. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Πέρα των ψηφοφοριών. Άρα τώρα μπορούμε να επανέλθουμε στο σημείο υπαριθμών 11 της Μεζής διατάξεως. Θα δώσω τώρα το λόγο ε, στον εισηγητή μας. Πρόκειται για πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας για τις δημοσιονομικές προοπτικές όσον αφορά το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο για το έργο ITER. Έχετε το λόγο εισηγητή. Die Πρόεδρε, όσον αφορά τις ε, προτάσεις για την ε, χρηματοδότηση του προγράμματος, είτε... σας παρακαλώ, λέει ο Κοιτάξτε, αυτά όλα συνδέονται με το πρόγραμμα Γαλιλαίος ε, και με τα συζήτηση για τα τρόφιμα των τελευταίων ετών. Τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο περίπλοκα. Στο ίτερ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ένα διεθνές πρόγραμμα όπου εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, Ιαπωνία, Νότιο Κορέα μεταξύ άλλων που συμμετέχουν και βέβαια δεν θέλω τώρα να αναφέρω με λεπτομέρειες ποιος θα δώσει ποια ποσά. Θα ήθελα μόνο να επισημάνω ότι η στάθμιση των ψήφων ακόμα και στα, ανάμεσα στα κράτη-μέλη ε, και την Κομισιόν, η στάθμιση πρέπει να αναθεωρηθεί ανάλογα ε, με το από πού προέρχονται τα κονδύλια. Κατά το παρελθόν, νομίζω ότι θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι κατά τη διάρκεια τη ε, Γερμανική Προεδρία μιλήσαμε για προγράμματα χρηματοδότηση σε σχέση με το πρόγραμμα ITER. Τώρα, η πρόταση που αντιμετωπίζουμε εδώ βασίζεται αφενός στις ε, αποφάσεις του Συμβουλίου της 12η Ιουλίου του 2010, όπου το Συμβούλιο ε, τοποθετήθηκε θετικά ε, σχετικά ε, με την ολοκληρωμένη και θετική ολοκλήρωση του προγράμματος είτε η Κομισιόν λοιπόν ενημερώθηκε για αυτή την πρόταση γιατί στις 27 και 28 Ιουλίου στο Κανταράς είχε συνεδριάσει η Επιτροπή που ασχολείται με το πρόγραμμα ΙΤΕΡ ε, και είχε γκρίνει σε γενικές γραμμές ε, αυτό το πρόγραμμα. Στη ανακοίνωση Κομισιόν αναφέρεται ότι όλα αυτά έγιναν με την επιφύλαξη ε, της περαιτέρω έγκρισης από την Επιτροπή Προπολογισμών. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ε, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα όπως και σε ορισμένους άλλους, σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή, Συζητάμε εδώ για το πώς ακριβώς πρέπει να χρηματοδοτούνται τα διεθνή προγράμματα, χωρίς όμως το Κοινοβούλιο να συμμετέχει, πόσο μάλλον να εισακούεται. Είτε πρόκειται για το πρόγραμμα σταθεροποίησης, είτε για άλλα εθνικά προγράμματα, πάντα αντιμετωπίζουμε το ίδιο μοντέλο. Τα πράγματα γίνονται πιο περίπλοκα, γιατί εδώ δεν πρόκειται απλά για αναθεώρηση του πολιτούς ε, χρηματοψηφιακού προγραμματισμού. Στην κατηγορία 2 μιλάμε για 400 εκατομμύρια, κατεβαίνει το πλαφόν, το ανώτατο όριο και αυτά τα 400 εκατομμύρια μεταφέρονται στο 2012 και το 2013 αυξάνοντας το ανώτατο όριο της κατηγορίας 1α και έχουμε να κάνουμε και με άλλες δόσεις και στοιχεία. Τα 460 εκατομμύρια βγαίνουν από το 7ο πρόγραμμα έρευσης, έρευνας και ανταυτού θα ε, εισέλθουν 100 εκατομμύρια το 2012 και ένα εξίσου σημαντικό ποσό το 2013. Θα θέλω λοιπόν να πω ότι η Επιτροπή Ήτρε ε, σε μία γνωμοδότησή της ε, καταφέρθηκε κατά αυτών των μεταφορών. Και άλλα 540 εκατομμύρια Μιλάμε για ένα σύνολο του 1,4 δις, άρα επανέρχομαι 540 εκατομμύρια θα οργανωθούν, λέει ο Μιλτή, θα διευκρινιστούν αργότερα. Και η Επιτροπή γράφει τα εξή. Στι διαβουλεύσει για τον προπολογισμό το Νοέμβριο του 2010 και εφόσον κρυφθεί απαραίτητο ε, στι ακόλουθε διαδικασίε ε, προπολογισμών που θα ακολουθήσουν, όπου πάντα συζητιώνται και εξαντλώνται οι δυνατότητε που υπάρχουν. Η Κομισιόν καλεί ε, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι τον συντονισμό του 2010 αυτή η δήλωσή της να ισχύει ως κοινή δήλωση. Και θέλω να πω ότι στο Συμβούλιο στη δική του τη δήλωση επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι ε, η συνεισφορά του Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 6,6 δις ε, μέχρι το 2016. Άρα δηλαδή αυτόματα εδώ μιλάμε για προγραμματισμούς και αριθμούς ε, οι οποίοι από το 2014 θα αρχίζουν να παίζουν κάποιο ρόλο. Όλα αυτά ε, γίνονται ακόμα πιο ενδιαφέροντα λόγω του ότι εμεί εδώ στο Κοινοβούλιο έχουμε μια διαφορετική άποψη για ένα τέτοιο πρόγραμμα. Κατά την άποψή μου, υπάρχει μια πολιτική ομάδα που διαφωνεί ριζικά ε, και εξ όσων γνωρίζω και στην Επιτροπή Έρευνας γίνεται μια συζήτηση όπου οτιδήποτε κουβεντιάζεται σε σχέση με το ίτερ θα πρέπει να συνεχίσει να χρηματοδοτείται ε, χωρίς ε, βέβαια να κινδυνέψει το πρόγραμμα, ε, καλύτερα να του ε, περικόψουμε λιγάκι ε, τις άκρες. Το λέω έτσι λαϊκά, όχι επιστημονικά, γιατί αυτά που περισσεύουν στις άκρες, όπως τα χαρακτήρισα, είναι εκείνα τα οποία κατ' ουσίαν δεν είναι επιστημονικά και για τα οποία μετά από αρκετά χρόνια θα γνωρίζουμε ποιε θα είναι οι επιπτώσεις τους στην πραγματική ενεργειακή πολιτική. Όλα αυτά λοιπόν τα γύρω-γύρω ε, μπορούν να περικοπούν γιατί δεν διευκολύνει την κατάσταση. Εξάλλου, η Κομισιόν είπε ότι μετά το 2013 θα υπάρχει ένα ετήσιο ε, κονδύλι ε, το οποίο θα προγραμματίζεται στις, στην επόμενη δημοσιονομική πρόβλεψη. Αυτά τα ξέρετε όλοι. Τώρα, στην έκθεση την διάμεση που υπάρχει ε, φύσεται ένα πρόβλημα, διότι με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνας υπερισχύει η ε, άποψη, η νομική άποψη ε, που προβλέπει την ομοφωνία. Βλέπουμε όμως ότι ε, σε περιπτώσεις που είναι κάτω από το 0,03% το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία. Εάν λοιπόν δεν μπορούμε να βρούμε κάποια ευελιξία ή κάποιες ε, άλλες μορφές αποθεμάτων για να χρηματοδηθούν τέτοιου προγράμματα, τότε πράγματι υφίσταται πρόβλημα και δεν ξέρω κατά πόσο η Κομισιόν μπορεί αυτό να το επιβεβαιώσει ή όχι. Εγώ ε, σε αυστριακές εφημερίδες γνωρίζω ότι όχι μόνο ο Υπουργός Γεωργίας αλλά και ο Υπουργό Οικονομικών, ο κύριος Πρόελ και οι δύο είπαν ότι αυτή τη μεταφορά κονδυλίων από την κατηγορία 2 στην κατηγορία 1α που θέλει η Κομισιόν διαφωνούν με αυτή τη μεταφορά. Νομίζω λοιπόν ότι εξάλλου ανοίγω παρένθεση αυτό αποδεικνύει ότι είχαμε δίκιο Όσον αφορά κάποιε διαδικασίε. είπαμε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει ευελιξία. Και εμείς ε, περιμένουμε την βελτιωμένη πρόταση τη Κομισιόν για την βελτιωμένη διοργανική συνεργασία με βάση τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι πρέπει να ξαναδούμε πολύ προσεκτικά το πρόγραμμα και να καταλήξουμε σε συνολική αξιολόγηση των κονδυλίων που πραγματικά είναι απαραίτητα. Αυτό είναι νομίζω ε, πολύ ενδιαφέρον με την έννοια ότι οι προτάσεις της Κομισιόν και του Συμβουλίου καταλήγουν στο ότι τελικά μιλάμε για το 2010 και κατά τα άλλα ε, η υπόλοιπη χρηματοδότηση θα λάβει χώρα το 2012, το 2013 και αργότερα με βάση την εμπειρία που ε, κάναμε με το πρόγραμμα Γαλιλαίος και το ε, πρόγραμμα για την οικονομική συγκυρία, αυτό κόστησε πάρα πολύ σε κόπο και χρόνο ε, και λόγω του ότι κατά τα επόμενα χρόνια θα έχουμε όλο και μικρότερα περιθώρια, εγώ Πραγματικά δεν πιστεύω ότι η Επιτροπή Προπολογισμών πρέπει να δεχθεί μια τέτοια πρόταση. Αλλά εμείς ε, πρέπει να περιμένουμε από την Κομισιόν, αφού εξετάσει εντελεχώς το σύνολο του προγράμματος, αν τελικά η Κομισιόν θεωρεί ότι πρέπει να συνεχιστεί ένα πρόγραμμα, μιλάμε για αυτό εδώ το ITER και λόγω του ότι έχει ε, σημασία για όλο τον κόσμο και το Κοινοβούλιο παίζει ε, καθοριστικό ρόλο, τότε η Κομισιόν να βρει μια σφαιρική προσέγγιση και όχι κάθε χρόνο να μας ε, καλεί να βρίσκουμε μια στιγμιαία προσέγγιση η οποία στη τελική ανάλυση αποβαίνει εις βάρος άλλων πολιτικών. Αυτή είναι μια δική μου πρόταση για να καταστήσει σαφές ε, στην Κομισιόν ότι με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούμε να έχουμε σοβαρή χρηματοδότηση του προγράμματος ITER. Εμείς περιμένουμε μια νέα πρόταση με ξεκάθαρο χρηματοδοτικό με ξεκάθαρη χρηματοδότηση και όχι να πρέπει συνεχώς να ασχολούμαστε με περικοπές και μεταφορές στις γραμμές προπολογισμού του 2012-2013. Κατά τα άλλα λοιπόν έχουμε κάποιο χρόνο, δεν πρέπει να δεχθούμε την πίεση της Κομισιόν απλά επειδή το Συμβούλιο αποφάσισε ότι τους επόμενους δύο μήνες θέλει να έχει μια συγκεκριμένη, ε, μια συγκεκριμένη προσφορά. Αυτό που ενδιαφέρει είναι ότι το αποτέλεσμα είναι καλύτερο από αυτό που έχουμε σήμερα στα χέρια μας. Ευχαριστώ κύριε Σιγητά. Πολλοί έχουν ζητήσει το λόγο και μετά θα δώσω το λόγο στον κύριο Γενικό Διευθυντή της Κομισιόν να μας πει τις απόψεις του και να απαντήσει και στις ερωτήσεις. Ο κύριος Αγγλούντ. Α, συγγνώμη. Ναι, James. Θα βοηθούσε να μιλήσει τώρα η Κομισιόν, να παρουσιάσει τις προτάσεις γιατί ακούσαμε την άποψη του Ράιμερ, παρά να μιλήσει τελευταία η Κομισιόν και να ακούσουμε τη θέση της τελευταία. Και εμείς να σχολιάσουμε και το 2 Μάλιστα, αν κατάλαβα καλά, ο Τζέιμς θέλει η Κομισιόν να πάρει τώρα το λόγο. Κύριε Γενική Διευθυντά, είστε έτοιμος, είστε έτοιμος Παρέμβατε. Président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 Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο για να σας αναφέρω την πρόταση της, ε, της να σας εκθέσω την πρόταση της Κομισιόν ε, και να υπογραμμίσω και εγώ την θέση μας σε σχέση με αυτά που είπε και ο εισηγητής. Ε, δεν θα πρέπει κανείς να αμφισβητήσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί στηρίζοντας το σχέδιο ΙΤΕΡ. Στο αυτό το σχέδιο βλέπουμε να υπάρχουν δυνατότητες ρύθμισης της του θέματος της ε, επάρκειας ενέργεια μακροπρόθεσμα. Και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση κέρδισε αυτό το σχέδιο, αυτό το πρόγραμμα μάλλον, ε, ενάντια στην υποψηφιότητα τότε της Ιαπωνίας. Όπως πολλά από αυτά τα προγράμματα, όπως και άλλοι τομείς που δεν έχουν διερευνηθεί, είναι δύσκολο να προβλεφθούν από οικονομικής άποψης με μεγάλη ακρίβεια. Από την άλλη πλευρά όλοι είμαστε πεπισμένοι ότι είναι πολύ σημαντικό να περιοριστούν και να ε, μετρηθούν τα κόστη, ακόμα και αν είμαστε σε τομείς όπου η τεχνολογία ακόμα δεν είναι απόλυτα καθορισμένη. Τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση Το επιπλέον κόστος που έχει εμφανιστεί και που τώρα έχει ανέλθει στο 1,4 δις για τη φάση κατασκευής μέχρι το 2020 έχει αποτελέσει αντικείμενο ανάλυσης και ελέγχου, οικονομικού ελέγχου καθώς και εξαιρετικά εις βάθος εξέτασης στο πλαίσιο του προγράμματος ITER αλλά και στο πλαίσιο του Συμβουλίου όπου εδρεύουν τα κράτη-μέλη. Mm. Οι όροι χρηματοδότηση μάλιστα έχουν αποτελέσει αντικείμενο ει βάθο συζήτηση στο πλαίσιο μια ειδική ομάδα που είχε δημιουργηθεί από την Ισπανική Προεδρία. Τα συμπεράσματα εκείνη τη ομάδα ήταν ότι όντω θα έπρεπε να προβλεφθεί μια χρηματοδότηση τη τάξη του 1,4 δις ευρώ για τα έτη 2012 και 2013 οι προτάσεις της Κομισιόν αποπειρώνται να βρουν ένα μέσο όρο ανάμεσα στην προσπάθεια που ζητάτε στο πλαίσιο του, που απαιτείται στο πλαίσιο του τίτλου 1α θα πρέπει να επιβληθεί αυτό και να γίνει εις βάρος άλλων προγραμμάτων που και αυτά ε, επιφέρουν ανάπτυξη και δημιουργούν απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη πλευρά την ανάγκη βεβαίως να μπορέσουμε να βρούμε χρήματα εντό εισαγωγικών φρέσκα, νοπά χρήματα εκεί όπου αυτά υπάρχουν. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο από τη μια πλευρά η Κομισιόν προτείνει μια αναδίπλωση 460 εκατομμύριων ευρώ στο εσωτερικό του τίτλου 1α, δηλαδή μέσα στο πρόγραμμα πλαίσιο, 100 το 2012 και 360 για το 2013, αφού εξετάσαμε την γεωργική κατάσταση το 2011, ξεκινήσαμε με βάση την υπόθεση ότι περίσευαν 400 εκατομμύρια που εύκολα μπορούσαν να κινητοποιηθούν και να μετακινηθούν από την τίτλο 2 στον τίτλο 1. Ξεκινάμε από την προϋπόθεση ότι τα 160 που περισσεύουν θα μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν Συγγνώμη, τα 560 περισσεύουν θα μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν με παρόμοιο τρόπο. Η μέθοδος αυτή, Προέδρε, αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή μέσω της ισχύουσας, με βάση μάλλον την ισχύουσα διοργανική συμφωνία. Δηλαδή, ανατρέχοντας στην ευελιξία του 0,03% του ΑΕΠ που μας επιτρέπει να πάρουμε μια απόφαση με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο. Τώρα βέβαια αυτό φαίνεται να αμφισβητείται από την νομική υπηρεσία του Συμβουλίου και να αποτελεί αντικείμενο μεγάλης αντίστασης από πλευράς των κρατών μελών. Υπάρχει εδώ δηλαδή, Πρόεδρε, μια στενή σύνδεση με την συζήτηση του θέματος της ευελιξίας στο πλαίσιο του κανονισμού που παρουσίασε η Κομισιόν μέσα στο πλαίσιο της εφαρμογής συνθήκης της Λισαβόνας. Τώρα, είναι επίγον ή όχι. Αυτό που θέλω να πω εγώ εδώ, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι η Κομισιόν έχει παρουσιάσει τη συμφωνία της, τη σύμφωνη της γνώμης όσον αφορά την baseline, δηλαδή για την ανάγκη χρηματοδότησης και τη μέθοδο χρηματοδότησης κατά τη διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου που συνήλθε τον Ιούνιο και δηλαδή αντρεφεράντουμ, δηλαδή υπό την προϋπόθεση της συμφωνίας της Δημοσιονομικής Αρχής, πιθανότατα προς τα τέλη του Σεπτεμβρίου θα γίνει μια νέα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕΡ και είναι σαφές πως οι εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα στραφούν προς εμάς και θα μας πούνε πώς εξελίσσεται η στάση της Δημοσιονομικής Αρχής στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την πλευρά της Κομισιόν θα Είμαστε ικανοποιημένοι αν μπορούσαμε να τους πούμε ότι οι εργασίες προχωρούν θετικά. Πράγμα που τουλάχιστον από την άποψη του Συμβουλίου, από την πλευρά του Συμβουλίου δεν ισχύει. Αλλά ελπίζω πως τουλάχιστον από την πλευρά του Κοινοβουλίου θα ισχύσει. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε κύριε Γενική Διευθυντία και δίνω το λόγο στους ε, βουλευτές μας, ο κύριος Χαγκλούντα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είχαμε μακρά συζήτηση για το θέμα αυτό στην ομάδα των φιλελευθερών πριν από κάποιε εβδομάδε και θα πρέπει να σα πω ότι είναι αρκετά σημαντικό το θέμα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Ράιμερ για τα πολλά και σημαντικά θέματα τα οποία ανέφερε. Εγώ προσωπικά δυσκολεύομαι πολύ. Ίσως επειδή είμαι σκανδιναβός ε, δεν καταλαβαίνω και πάρα πολύ καλά πώς είναι δύσκολο να μπορέσει κανείς ε, να ανταποκριθεί σε ένα προϋπολογισμό ε, από τη στιγμή που έχει και κάτι τεράστια περιθώρια εκτός και αν έχει γίνει τελείως λάθος σχεδιασμός και πραγματικά δεν ε, με πείθεται καθόλου λέγοντας ότι δεν είναι εύκολο να γίνουν προβλέψεις σε ένα τέτοιο τομέα ερευνητικό και τέτοια δεν στέκει αυτή η εξήγηση γενικά οι εξηγήσει για το, οι αιτιολογήσεις μάλλον για το γιατί καταλήξαμε σε αυτή την κατάσταση δεν ισχύουν, δεν στέκουν. Είναι εν γέννη εύκολο να υιοθετήσει κανεί την προσέγγιση του εισηγητή μα και θέλω να επιστήσω την προσοχή σα στο γεγονό ότι τώρα προτείνουμε να πάρουμε πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ από το FP7, δηλαδή από το πλαίσιο, πρόγραμμα πλαίσιο 7. Τεράστιο ποσό. Και αν θέλετε να τα πάρετε από την έρευνα και την καινοτομία, δεν νομίζω ότι μπορούμε να τα πάρουμε όλα αυτά τα χρήματα από την έρευνα. Ξέρω ότι και αυτό έρευνα είναι, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα σημαντικά ερευνητικά προγράμματα στην Ευρώπη. Και το να πάρουμε τόσα πολλά χρήματα και να τα βάλουμε μόνο σε ένα, ε, νομίζω θα μας ε, θα μας θέσει στην ίδια κατάσταση όπως είμαστε με το 2020, τη στρατηγική του 2020. Ας μην καταλήξουμε λοιπόν και εδώ λαμβάνοντας τις λάθος αποφάσεις. Ε, όπως με τη συνθήκη της Λισαβόνας, συστηρίζω τα όσα προτείνει ο Ράιμερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην Επιτροπή Ενέργειας και Έρευνα συζητήσαμε διαμακρών για το θέμα αυτό. Για μας ε, το πρόγραμμα ΙΤΡΕ είναι ένα θεμελιώδες ε, πρόγραμμα βάσης, ε, το οποίο βέβαια ξεκινήσει εδώ για πολλά χρόνια και θα διαρκέσει εξίσου πολλά στο μέλλον. Είναι λοιπόν σημαντικό κατά την αναδιοργάνωση και τον ε, εξορθολογισμό του προγράμματος να ορίσουμε νέα ορόσημα. Δηλαδή το τι μπορεί να γίνει πολύ συγκεκριμένα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον. Τώρα, όσον αφορά τις ε, τροπολογίες της Κομισιόν και του Συμβουλίου, ε, στο πλαίσιο του 7ου προγράμματος πλαίσιο του αποκαλούμενου CHIPS, ή στο πλαίσιο της γεωργίας όπου θέλουμε να προάγουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, νομίζουμε ότι εκεί δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν περικοπές. Ειδικά ε, λόγω της ε, χρηματοπιστωτικής κρίσης, οι αριθμοί του 2010 θα πρέπει να ισχύσουν και για το 2011. Χρειαζόμαστε λοιπόν τη συνέχεια. Και βεβαίω, αν το κατάσταση βελτιωθεί, αν σταθεροποιηθεί, ε, ίσως από το 2014 το πρόγραμμα πλαίσιο να μπορεί να πρικοδοτηθεί με φρέσκο χρήμα. Ε, ίσως ε, μπορούμε να ξανασυζητήσουμε και το πρόγραμμα για το διοξίδιο του άνθρακα που ασχοληθήκαμε τόσο πολύ με αυτό. Εκεί δεν υπάρχει δέσμευση του Συμβουλίου. Από τα τέλη για το διοξίδιο του άνθρακα θα μπορούμε να βρούμε αυτό το φρέσκο χρήμα, αλλά σίγουρα όχι από τα υπάρχοντα ε, προγράμματα. να περικόψουμε την γραμμή 20 κατά τη γραμμή κατά 20% αυτό νομίζω ε, για μας είναι απαράδεκτο. Γκόρια Χάμπερ. Sí, gracias, Presidente. Muy brevemente, porque creo que estamos bastante de acuerdo con... Κύριε Πρόεδρε, σε γενικές ε, γραμμές ε, συμφωνούμε με αυτά που μας είπε ο συγητής, αλλά θέλω να πω το εξής. Τώρα, αυτή τη στιγμή, βλέπουμε ενδεικτικά ένα παράδειγμα προς αποφυγή όσον αφορά τις προετοιμασίες φροντικές που διακρίνονται από τόση λιτότητα και, και, και αυστηρή πολιτική, γι' αυτό και κατά τη γνώμη μας αυτό είναι απαράδεκτο. Πρώτα-πρώτα βέβαια θα πρέπει τα 400 εκατομμύρια να δούμε τι θα κάνουμε γιατί πρόκειται για τη συγκεκριμένη τεχνική που βάζουμε σε ε, σε τέτοιε αγγείλε τα 400 εκατομμύρια είναι μια τεχνική του Συμβουλίου που θα πρέπει να δούμε κατά πόσον ε, είναι κάτι το ε, που το δεχόμαστε ή όχι, αλλά, αλλά δεν είναι δυνατόν να τα αφαιρέσουμε από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Αυτό το οποίο είναι δυνατόν να γίνει είναι να θέσουμε τις προτεραιότητες και όταν ε, βάζουμε αυτά σε κάποιο σαν αποθεματικό και αν χρειαστεί τα παίρνω από εκεί γιατί πρόκειται για κάποιες πάρα πολύ σημαντικές προτεραιότητες που έχουμε εδώ πέρα κατόπιν έχουμε τα 540 εκατομμύρια ε, που αφορούν την χρηματοδότηση και αυτό το έκαναν με μία παρόμοια μέθοδο. Άρα χρειάζεται μία καινούργια πρόταση. Και επίσης θα πρέπει να συνεχίσουμε ε, τον αγώνα μας για να υπάρχει περισσότερο περιθώριο ελιγμών, περισσότερη ευελιγμία στον προπολογισμό για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές Άρα θα πρέπει να συνεχίσουμε τον προβληματισμό για τα θέματα αυτά, γιατί ποτέ δεν εξαντλείται ο προβληματισμός. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Τώρα έχουμε μια άλλη φωνή από την Ισπανία. Ο ίδιος ο Σαλδόρ Γκαρίγα. Ε, εγώ θα είμαι ακόμα πιο σύντομος, Πρόεδρε. Έχουμε αυτό το οποίο μας ζητούν. Είναι ότι θα πρέπει να πουλήσουμε τα παπούσια για να αγοράσουμε το, το καπέλο. Ε, Επομένω, βλέπουμε ότι αυτό είναι φινησιγενές σαν, σαν πρόταση ε, Και μας ζητείτε να σας πούμε αν συμφωνούμε. Το ίτερ είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα χρειαζόταν διπλάσια ή τριπλάσια πρικοδότηση από την κοινότητα. Αυτό μας βρίσκει όλους σύμφωνους. Πρόκειται για ένα μεγάλο όραμα, πρόγραμμα για το μέλλον την αλλαγή του κλίματος, για την μετανολική ανάπτυξη, για την ενέργεια, οπότε έτσι, υπ' αυτού τους όρους, όχι. Όπως είπε και, η συνάδελφος Χάιντερ, ε, να παίρνουμε χρήματα πρόγραμμα πλαίσιο, να αφήνουμε τη μισή χρηματοδότηση να εκρεμεί και να ελπίσουμε ότι θα προγύψει κάποια υπέροχη λύση στους επόμενους προϋπολογισμούς. Αυτό δεν είναι δημοσιονομικός προγραμματισμός και θα πρέπει όπως πάντοτε ε, να, να, να, να σπεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εις βοήθεια του Συμβουλίου για να έχουμε ε, κάποιες ε, λύσεις οι οποίες θα ευρεθούν στο γόνατο και χωρίς να λεφθεί υπόψη το πολιετές πρόγραμμα. Οπότε ε, θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα γιατί δεν έχει ληφθεί υπόψη η ενδιάμεση αναθεώρηση. Ούτε καν γνωρίζουμε αν υπάρχει κάποιο είδου αξιολόγηση, δεν έχουμε αριθμητικά στοιχεία σε σχέση με το πώ γίνεται η εκτέλεση των πολιωτών προγραμμάτων για τη συγκεκριμένη περίοδο των δημοσιονομικών προοπτικών υπ' αυτού, του όρου. Επομένω, το Κοινοβούλιο δεν είναι δυνατόν να πει ναι σε αυτή την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι αλήθεια ότι έγινε εδώ απόπειρα να γίνουν οικονομίες από εκεί που δεν γίνεται. Όμως μια τέτοια πρόταση είναι απαράδεκτη άρα θα πρέπει να διαβιβαστεί ή στο Συμβούλιο ότι θα πρέπει ή να περιμένουμε την μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση των σημερινών προοπτικών ή θα πρέπει το ζήτημα της χρηματοδότησης Twitter να μπουν στις επόμενες προοπτικές γιατί σήμερα όπως έχουν τα πράγματα δεν εξυπηρετούν. Τώρα έχουμε και άλλους ε, συναδέλφους που έχουν ζητήσει το λόγο από ό,τι βλέπω έχει διαμορφωθεί μία συνένεση και γι' αυτό νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε γρήγορα. Η κυρία Ιζαμπέλ Ντιρόν ζητεί τώρα το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη στα πλαίσια αυτών των συγκρίσεων. Θα πρέπει να ξέρετε ότι εμείς καταρχήν είμαστε κατά του ίτερος πράσινοι. Από την άλλη μεριά όμως θα πρέπει να δούμε τα επιμέρους κομμάτια του ψηφιδωτού, του μοσαϊκού και βλέπουμε ότι η αντιμετώπιση τώρα δεν είναι σοβαρή. Έχουμε τη νέα Κομισιόν και για τις ε, δημοσιοποιείς προοπτικές είχαν πει ότι θα χρηματοδοτήσουν της, ε, την πολιτική ενόψη του 2020 και τη φυγή προς τα εμπρός και στα πλαίσια του Ίτερ αυτά δεν γίνονται. Και δεν είναι σωστό να το συγκρίνουμε με τον Γαλιλαίο που είναι χρήσιμο, ενδιαφέρον για πάρα πολλούς ως πρόγραμμα. Αυτά επί τη ουσία. προτιμούν το Γαλλίο από το Ήτρε. όμω, όσον αφορά τη μέθοδο και τη μεθοδολογία θεωρώ όπω και άλλοι συνάδελφοι ότι αυτό που μας προτείνουν είναι απαράδεκτο. Η κατάσταση αυτή είναι αφόρητη. Δεν είναι δυνατόν έτσι να καθορίζουμε τις ε, δημοσιονομικές μας προτεραιότητες. Δηλαδή... Πρόεδρε, Θέλω να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο συγητής. Όμως ε, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση προς την Επιτροπή. Διότι αυτά που συζητάμε σήμερα προβλέπουν ότι το 2010 από την ε, στήλη 2 ε, θα αφαιρεθούν 400 εκατομμύρια ευρώ. Και έχουμε ένα άλλο σημείο, το 24, στη μέση διάταξη για την ε, έγκαιρη προειδοποίηση όπου βλέπουμε ότι το 2010 τους πρώτους τέσσερις μήνες εκτέλεσης αυτού του προπολογισμού κατ' ουσίαν έχουμε μικρότερες δαπάνες σε σχέση με τις προβλέψεις, ε, περίπου των 200 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά που είχαν σχέση με την αγορά. Όμως, ανταυτού, αύξηση δαπανών για άμεση ενισχύσεις της τάξης των 328 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Άρα δηλαδή, σε σχέση με αυτά που μας λέει η Κομισιόν, έχουμε ε, αύξηση των δαπανών, είναι μεγαλύτερο το ποσό της αύξησης, ε, κατόπιν τούτου, εγώ θεωρώ ότι εδώ έχουμε μία αντίφαση. Από τη μια έχουμε μία ανακοίνωση ότι δεν πανάμε περισσότερα χρήματα σε σχέση με αυτά που έχουμε προβλέψει και από την άλλη έχουμε ε, μία ε, πρόβλεψη 400, μείωση 400 εκατομμύριων ευρώ, αφαίρεση αυτού του ποσού για να χρηματοδοτηθεί το πρόγραμμα ITER. Η κυρία Γκρέσλε έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα ήθελα να πω ότι ένα πράγμα εντυπωσιάζει, ότι η διαχείριση των μεγάλων προγραμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ε, μη ικανοποιητική. Αν δούμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα, τότε θα καταλήξουμε στο ότι ε, δεν θα πρέπει να ε, ασχολούμεθα με τα δημοσιονομικά αν δεν προβαίνουμε και σε διαρθρωτικές αλλαγές. Αυτό εδώ το βλέπουμε στο πρόγραμμα ITER. Η Επιτροπή Προπολογισμών το 2008 έκανε μια μελέτη όπου αναλύει το πρόγραμμα Γαλιλαίος ε, και το ITER ε, από, κυρίως σε σχέση με το ΣΕΠΤ. Αυτή λοιπόν η μελέτη είναι πολύ σημαντική. Δείχνει ποιο είναι, ποιο είναι το management που έχουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δει σε βάθος ε, τις δομές του Ε, Βαρκελόνη, Εκεί, παραδείγματο χάρη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει το 45% των χρημάτων, αλλά δεν έχει σχεδόν καθόλου φωνή. Άρα, δηλαδή, αυτό ε, που χρηματοδοτεί ε, θα πρέπει και κατά κάποιον τρόπο να ορίζει τι θα συμβαίνει. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να συστήσουμε ένα δεύτερο συμβούλιο το οποίο ε, θα φωτίσει αυτή την ε, τόσο ε, περίπλοκη τεχνολογία. Γιατί τέτοιου καταστάσεις καταστάσει θα τις βιώσουμε επανειλημμένα. Και εφόσον υπάρχουν χρήματα, ή αν θέλετε να διαθέσουμε χρήματα, μόνο εφόσον υπάρξουν διαρθρωτικές αλλαγές. Και τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο James Ellis έχει το λόγο. Εγώ θα πω κάτι διαφορετικό από τους υπολείπους. Εγώ στην περιφέρειά μου ασχολούμαστε ε, ιδιαίτερα με την σύνδεξη και ήμουν ιδιαίτερα φιλελε... Ε, περήφανος ανέκαθεν ε, που ανέκαθεν παίξαμε σημαντικό ρόλο για την πρόθεση της ε, σύνδεξης, ενώ οι πράσινοι και άλλοι που αποτίθεται ότι είναι πιο προοδευτικοί το έχουν ε, αφήσει. Πρόκειται για ένα παγκόσμιο πρόγραμμα, φαίνεται, τυχαίνει να βρίσκεται ε, στη Ένωση και μάλιστα στη χώρα σας, Πρόεδρε, και γι' αυτό θα προσέξουμε, θα πρέπει να προσέξουμε πριν πούμε ότι δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση. Έχει, είναι σοβαρό πρόβλημα, έχει σοβαρά, μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζει, αλλά ε, θα πρέπει ίσως αυτοί οι άνθρωποι που το διαχειρίζονται να έρθουν να μας πούν ε, τι, τι, τι ακριβώς γίνεται. Ε, παρά να το απομακρύνουμε και να το απορρίπτουμε κατευθείαν. Το ερώτημά μου στο τέλος είναι ότι αν η Επιτροπή ε, ακολουθήσει την Συμβουλή να ζητήσει μια άλλη πρόταση και να το βάλουμε στη μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική αναθεώρηση, όλοι ξέρουμε ότι αυτό θα γίνει μετά από το 2013. Τι σημαίνει αυτό, ότι το πρόγραμμα θα σταματήσει να υπάρχει, γιατί τότε αναλαμβάνουμε την ευθύνη για το όρομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για το ρόλο της σε παγκόσμιο επίπεδο. Φαίνεται να είμαστε κάπως εσωστροφείς όταν εξετάζουμε τα συστήματα ασφάλεια ασφάλειας ε, ανεφοδιασμού ενέργεια. Η σύνδεξη νομίζω πως είναι ένα από, αυτά τα, από αυτές τις λύσεις. Η Κομισιόν λοιπόν θα μας πει ακριβώς ναι, πού ναι. βρισκόμαστε. Ευχαριστώ, James. Όντω, αφού το Βρετανικό Συντηρητικό Κόμμα είναι υπέρ του προγράμματος πρέπει να το ξανασκεφτούμε μια δεύτερη φορά πριν διατηρήσουμε αυτή την εχθρική στάση. Τέσσερι ακόμα έχουν ζητήσει το λόγο και κλείνω το κατάλογο των ομιλητών γιατί έχουμε πολύ πολύ φορτωμένη μερίσια διάταξη. Πήγα να βιαστώ και να πω ότι υπάρχει συνένεση, αλλά όχι. Είναι διχασμένες οι απόψει. Κύριε Καρβάλιο, σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να πω πως θεωρώ το ΙΤΡΕΝ πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, γιατί είναι το πρώτο παγκόσμιο πρόγραμμα τέτοιων διαστάσεων, εδρεύει στην Ευρώπη και εγώ πιστεύω πως η σύνδεξη είναι πολύ σημαντικό ζήτημα για το μέλλον της Ευρώπης και επίσης θεωρώ ότι η ευελιξία στην έρευνα είναι πάρα πολύ σημαντική. Ο, τούτων λεχθέντων όμως, ε, αν κανείς εξετάσει το πρόγραμμα ITER, βλέπει πως δεν είναι μόνο θέμα ευελιξίας και έρευνας, είναι ακόμα πολύ νωρίς στο πρόγραμμα για να οφείλεται αυτή η ανάγκη νέας χρηματοδότησης σε νέα ευρήματα. Όχι, νομίζω πως ε, πρόβλημα υπάρχει στην ε, βέλτιστη χρήση της δομής. Και συμφωνώ με τον συνάδελφο Γκρέσλε ότι θα πρέπει να εξετάσουμε την δομή και τη διαχείριση του προγράμματος. Γιατί από τη μια πλευρά, ναι, δεν πρέπει να το σταματήσουμε, αλλά δεν κάνουμε και τίποτα στη δομή του, για να αλλάξει η δομή του, αυτό θα συμβεί ξανά και ξανά. Πρέπει λοιπόν να θέσουμε κάποιους όρους, να εξετάσουμε πολύ καλά πώς λειτουργεί το ΙΤΕΡ, γιατί συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν. Να καταλάβουμε, να έχουμε πιο βαθιά κατανόηση του τι συμβαίνει και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε τέτοιου είδους καταστάσεις να μην ξανά συμβούν. Υποστηρίζω λοιπόν το ότι θα πρέπει να καταλάβουμε ακριβώ τι συμβαίνει για να μπορέσουμε να αποφασίσουμε. Ευχαριστώ. Ο κ. και Μπράντι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ πιστεύω ότι το πρόγραμμα ITER είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει μέγα μέλλον μπροστά του. Είμαι πεπισμένος περί αυτού. Ωστόσο υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Δεν πρέπει να αναμειχνύουμε το μέλλον του προγράμματος με τα διαδικαστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εδώ. Εγώ θα ήθελα να τα χωρίσουμε αυτά, να τα ξεχωρίσουμε. Έχω μια ερώτηση προς την Κομισιόν. Αυτό είναι, είπαμε, διεθνές πρόγραμμα. Νομίζω συμμετέχουν, είπα, η Ιαπωνία, χώρες, οι συνεργάτες. Ε, θα πρέπει να είμαστε περήφανοι που εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση μπορέσαμε να, έχουμε αυτό το να κρατήσουμε το πρόγραμμα αυτό εδώ στην Ευρώπη και όχι σε μια από τις άλλες αυτές χώρες. Το θέμα είναι αυτό το 1,5 εκατομμύριο που μας λείπει μέχρι το 2020. Είναι μόνο το ευρωπαϊκό κομμάτι του επιπλέον κόστους είναι το σύνολο του πρόσθετου στόχου για το οποίο πληρώνουμε εμείς οι Ευρωπαίοι. Δηλαδή υπάρχουν δυνατότητες οι άλλες χώρες να βάλουν και αυτές κάτι τι. Να καλύψουν κάποιο μέρος αυτού του επιπλέον κόστους. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Ο κύριος Σούριαν. Ευχαριστώ πρόεδρε και συμφωνώ ότι θα πρέπει να κάνουμε κάτι στα σοβαρά διότι συμφωνώ με τον Κλοντ. Και επίσης, μια που ήμουν εισηγητής στον προπολισμό της χρήσης του 2010, εγώ δεν μπορώ να είμαι υπέρ τέτοιων μεθόδων, τέτοιων λύσεων. Και αυτό το οποίο θεωρώ είναι ότι, όπως είπε εσείς πρόεδρε, Καταρχήν υπάρχει εδώ θέμα μια που δεν μπορούμε να δεχθούμε τέτοιες μεθόδους. Και να δούμε η περισσότερη από μας εάν επιμένουμε στη θέση μας. Μιλάμε για 1,4 δις ευρώ. Αυτό είναι το, το, το κόστος το οποίο περισσεύει και αυτό που δεν μπορούμε να δεχθούμε είναι να συμφωνήσουμε με λύσεις τέτοιες που για να λυθεί ένα καινούριο πρόβλημα ξανανοίγουν ένα παλιό το οποίο είχε κλείσει. Η κυρία Γέννης το λόγο, είναι τελευταία ομιλήτρια. Κύριε Πρόεδρε, στη δική μου την πολιτική ομάδα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το πρόγραμμα ITER. Εγώ ανήκω στους ε, ενθουσιώδεις ε, όπως και ο κύριος Αρλής, ε, το βρίσκω ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό πρόγραμμα Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ισχυρή θέση όχι μόνο ως Βρετανία αλλά και ως Ευρώπη. Και αυτό θα πρέπει να είναι ο στόχος μας. Αυτά ως προς το πρόγραμμα. Πάμε τώρα στη χρηματοδότηση. Νομίζω ότι είναι παντελώ απαράδεκτο το ότι ε, αναφέρουμε μια το ένα, μια το άλλο, ε, τι μπορεί, τι δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί, όπου το Συμβούλιο και ο Κομισιόν ε, μας πιέζουν και λένε ότι ε, πρέπει να δεχτείτε περικοπές σε άλλους τομείς για να χρηματοδοτηθεί το πρόγραμμα αυτό. Τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα. Ε, χρειαζόμαστε λοιπόν καταρχήν αναθεώρηση του μέσοπρόθεσμου, της μέσοπρόθεσμης χρηματοδότησης και ελπίζω να κατατεθεί σύντομα μία πρόταση για να μπορούμε να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες χρηματοδότησης και να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες και για νέα προγράμματα ε, ίσως ε, το πρόγραμμα είτε επιπρόσθετα κονδύλια για το πρόγραμμα Γαλιλαίος και οτιδήποτε άλλο προκύπτει από τη συνθήκη της ε, Λισαβόνας. Γιατί αλλιώς ε, τελικά ε, δεν θα νιώθουμε ότι έχουμε σταθερό έδαφος κάτω από τα πόδια μας. Θα ζητήσω από το Ράιμερ να βγάλει τα συμπεράσματα και να μας πει Ποιε είναι οι πλέον πληροφορίες που θέλει να ζητήσει από την Κομισιόν και η Κομισιόν θα, θα το τις δώσει είτε προφορικά είτε γραπτά. Αλλά θα ήθελα και εγώ να κάνω μια παρατήρηση. Καταρχήν, είναι κάπως παράξενο να βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μάλιστα υπό την πίεση του Συμβουλίου αρνήθηκε μέχρι στιγμή να θέσει επιτάπωση μία πρόταση αναθεώρηση των ισχυούσων δημοσιονομικών προοπτικών, εκτό ξαφνικά για ένα μόνο πρόγραμμα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει, όλοι, δεν το υποστηρίζουν όλοι στην Επιτροπή, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια ε, πλειοψηφία που είναι υπέρ αυτού του προγράμματο, το οποίο είναι αξιόλογο και που δεν υπάρχουν αρκετά προγράμματα τέτοιου μεγέθου παγκοσμίου ε, εμβέλειας, όπου μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει και την ε, πρωτοκαθεδρία. Ας, ταυτόχρονα όμως είναι και δύσκολο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητά, που, που του ζητούν μια αναθεώρηση δημοσιονομικών προοπτικών, να, μάλλον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητά αναθεώρηση δημοσιονομικών προοπτικών για τη Λισαβόνα, και να το, το αρνείται το Συμβούλιο και γίνονται μάλιστα και αναφορές για μια στάση που μπορεί να θεωρηθεί ανεύθυνη του Κοινοβουλίου που θέλει να κάνει δαπάνες και να τροποποιήσει τις οροφές και ταυτόχρονα μόλις υπέρχεται ένα θέμα που είναι σημαντικό για το Συμβούλιο και την Κομισιόν να δέχονται όχι να, όχι να ανεβάζουν τις οροφές αλλά μπας περιπτώσει να ανακατανείμουν τα χρήματα. Ε, είναι πολιτικό το ζήτημα και σας το τονίζω. Δεν είναι ίσονο σημασία μάλιστα. Αυτό που είναι βέβαια διασκεδαστικό σε αυτή την παρουσίαση είναι ότι λέει μηδέν για το 2011 και οι πρώτες επιπλέον δαπάνες θα ξεκινήσουν το 2012. Γιατί λοιπόν να μην περιμένουμε το 2012. Γιατί όχι, θέλουν να πάρουν μάλλον 400 εκατομμύρια από το γεωργικό προπολογισμό του 2010. Μα βλέπουμε ποιο είναι ο πειρασμό και πρέπει ω ε, Επιτροπή Προπολογισμού να τα συζητήσουμε μεταξύ μα. Γιατί αν αυτά τα 400 εκατομμύρια δεν τα πάρουμε τώρα, μπορεί να αποτελέσουν πλεονάσματα εκτέλεσης στο τέλος του έτους υπό την ε, επιφύλαξη της αναθεώρησης που, που ζητάει ο κύριος ε, Ραβίδη. Άρα λοιπόν, θα μπορούσαμε να κρατήσουμε για μια ευρωπαϊκή πολιτική πλεονάσματα, αυτό είναι το δόλωμα της Κομισιόν, που διαφορετικά θα σταλούν πίσω στα κάτι μελη Πρέπει να πούμε όχι δηλαδή, μήπως πρέπει να το ξανασκεφτούμε. Δυστυχώς όμως για την πρόταση τούτη διαπιστώνω, ακούγοντα τα μέλη, ότι αυτοί που συμπαθούν την δαπάνη, δεν συμπαθούν το, τα έσοδα ενώ και, και Δύσκολο να δούμε ποια θα είναι η πλειοψηφία. Κύριε Σιγητά, μήπως θέλετε εσείς τώρα να συνοψίσετε. Κοιτάξτε, καταρχήν ε, να πω ότι συμφωνώ με αυτά που είπε ο Πρόεδρος ε, και αυτό που είπε και ο συνάδελφος ε, προηγουμένως σε σχέση με τις συνεισφορές όλων των άλλων συμμετεχουσών χωρών και εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικό να ε, αποκτήσουμε περισσότερες ε, πληροφορίες ε, για όσα κράτη συμμετέχουν στο πρόγραμμα ITER. Αυτά που συζητάμε εδώ δεν είναι διαδικαστικά. Πρέπει να το πούμε αυτό. Η τεχνική για τον προπολογισμό κατ' ουσίαν είναι πάντα έντονα πολιτική. Συμφωνώ με αυτά που είπε η συνάδελφος κυρία Καβάλιο σε σχέση με το σύνολο του προγράμματος. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι όλα αυτά που μας είπε ο κύριος Έλλης, οι παραδοχές του, ευσταθούν. Και έχω την εντύπωση ότι οι περισσότεροι πιστεύουν ότι το ίτερ είναι ένα πρόγραμμα που χρήζει στήριξης και ότι ειδικά όσον αφορά το πρόγραμμα αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στην πρωτοπορία. Αν όμως ισχύουν όλα αυτά τότε θα πρέπει και η Κομισιόν και το Συμβούλιο να γνωρίζουν τις δυσκολίες και να υποβάλουν μια διαφορετική πρόταση έτσι ώστε το πρόγραμμα ITER κατά τα επόμενα χρόνια να είναι πάνω σε σταθερά πόδια και όχι αυτή την πολιτική του σταγονόμετρου όπου αναγκαζόμαστε κάθε χρόνο, ανά δύο-τρεις μήνες να έχουμε διαπραγματεύσει. Μα τι είδου ε, αξιοπιστία είναι αυτή να μιλάμε κάθε φορά για 45 εκατομμύρια. Γελιοποιούμαστε με τον τρόπο αυτό. Γι' αυτό λοιπόν να πω στο Γενικό ε, Διευθυντή ότι ε, τέλη Σεπτεμβρίου θα υπάρξει κάποιο συμβούλιο για το ΊΤΕΡ. Εκεί λοιπόν το Κοινοβούλιο θα πρέπει να αντιδράσει λιγάκι θετικότερα από ό,τι έχει συμβεί μέχρι τώρα. Και όλα αυτά που λέει το Συμβούλιο ε, θα έπρεπε να τα έχει σκεφτεί νωρίτερα. Πάντως ε, η δική μου άποψη είναι ότι εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση με βάση μια τροποποιημένη και βελτιωμένη πρόταση. Βεβαίως ε, το Νοέμβρη να κάτσουμε όλοι σε ένα τραπέζι και να προσπαθήσουμε μέσα από τις διαπραγματεύσεις, να βρούμε μια καλή λύση. Αλλά, σας λέω, λαμβάνοντας υπόψη αυτά που ελέγχθησαν σήμερα εδώ. Και μπορείτε να θεωρήσετε ότι αυτό που σας είπα είναι η πρώτη άποψη της Επιτροπής Ευρωεκολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όχι όμως ε, να λέμε 400 εκατομμύρια από την ε, κατηγορία 2 και μετά ε, να ξεκινήσει το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο με όλες τις σχολείς που έχει. Μην ξεχνάτε ότι εδώ στο Κοινοβούλιο χρειαζόμαστε τις πλειοψηφίες και αν μία πρόταση τελικά δεν εφαρμοστεί, δεν θα υπάρξει και πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο και τότε η καταστροφή θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Γι' αυτό λοιπόν λέω στην Κομισιόν να καταθέσει μια νέα πρόταση και με βάση αυτή την αναθεωρημένη πρόταση θα δεχθούμε τις διαπραγματεύσεις. Ο Αλλά έχει δίκιο. Τώρα ε, στο ε, προϋπολογισμό δεν προβλέπεται τίποτα για το 2011 αλλά ε, τα χρήματα του 2010 υποτίθεται θα μεταφερθούν στο 2011 και στο 2012. Τα άλλα θέματα όμως παραμένουν ανοιχτά. Νομίζω λοιπόν κύριε Πρόεδρε ότι μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση, να πούμε ότι συμφωνούμε όλοι ότι η Κομισιόν πρέπει να καταθέσει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για το ε, σύνολο της ε, περίοδου χρηματοδότησης. Δεν πρόκειται εδώ μόνο, μόνο για το πρόγραμμα ITER. Εκεί να αναζητηθούν οι λύσεις ή τουλάχιστον να προετοιμαστούν οι λύσεις έχοντας κατά νου ε, τον συντονισμό του Νοεμβρίου. Τότε όμως τα πράγματα να είναι πιο ρεαλιστικά, πολύ καλύτερα από αυτά που μας έχει προτείνει σήμερα και η Κομισιόν και το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Κύριε Διευθυντά. Ευχαριστώ κύριε εισηγητά και θα συνεχίσουμε όπως μας πρότεινε ο εισηγητής μας. Σημείο 12 της ημερήσιας διάταξης πρόκειται για μια ανταλλαγή απόψεων για την έκθεση της κυρίας Αντρέσεν για την βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης και του πλαισίου σταθερότητας της Ένωσης, ειδικότερα στη ζώνη του ευρώ. Κυρία εισηγήτρια, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι αυτό που τώρα συζητούμε είναι το πώς θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε την, ε, το σύμφωνο σταθερότητος και ανάπτυξης. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Και έχουμε και τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ορίζει στο άρθρο 126 κάποιες ε, διαδικασίες που προβλέπονται σε περίπτωση παραβάσεων. Όμως αυτό δεν έχει θεσπιστεί για το σύμφωνο σταθερότητα και ούτε καν επιλαμβάνεται τέτοιων περιπτώσεων το δικαστήριο του Λουξεμβούργου. Θα πρέπει να δούμε μας τι κυρίως μπορεί να υπάρξουν για να δούμε τι θα γίνει με τις ε, ε, προσπάθειές μας ε, για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση από μια άλλη κρίση. Προβλέπονται οι διαδικασίες, όμως θα πρέπει να τις εφαρμόσουμε. Και γι' αυτό και ε, νομίζω ότι θα πρέπει το Συμβούλιο να αναλάβει δράση. Η δεύτερη πτυχή που τώρα θα ε, έχει να κάνει με αυτή μας την προσπάθεια είναι το κατά πόσον θα μπορέσουμε να εμπλέξουμε τα εθνικά κοινοβούλια διότι είναι εις καλύτερα να μπορέσουν να επισημάνουν τα ορθότερα μέτρα και να εγγυηθούν την ε, εκτέλεσή τους. Ο πλευράς προϋπολογισμού και του μηχανισμού σταθεροποίησης θα πρέπει να θυμόμαστε ότι οι εγγυητές αυτού του παγιού του 260 είναι τα κράτη-μέλη πολλά των οποίων επίσης υφίστανται κρίση. Άρα θα ήθελα να μου πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποιε είναι οι επιπτώσει όσον αφορά την πιστοληπτική ικανότητα και την αξιολόγησή τη. Τι γίνεται όσον αφορά αυτέ τι δαπάνε από το προπολογισμό, αν κληθούμε να τιμήσουμε τη δεσμευσή μα για αυτή την εγγύηση. Ευχαριστούμε κυρία εισηγήτρια, η κυρία Ανδρέασεν. Έχει αυτή την περιεκτική και σύντομη έκθεση που μας παρουσίασε. Έχετε το λόγο τώρα. Και εγώ θα είμαι σύντομος, λέει ο μια ματιά στις προτάσεις Ανδρέας Δυστυχώς, αντιβαίνουν στις δικές μας απόψεις. για το σύμφωνο σταθερότητας και για τον καινούριο μηχανισμό χρηματοοικονομικής σταθερότητας. Εμείς δεν θα εγκρίνουμε αυτή την έκθεση και θα δούμε σε μεσόμενες μέρες αν θα προβάλλουμε τροπολογίες ή αν απλώς θα καταψηφίσουμε. Ο επόμενος συνάδελφος είναι ο κύριος Γκαρίγα. Μάλιστα, πρόεδρε. Χωρίς να φτάσω στο σημείο να σας πω αυτά που ο κύριος Φάρμ, εγώ θεωρώ ότι στο σημείο υπαριθμών 1 ότι δεν είναι αρμοδιότης της Επιτροπής των Προπολογισμών να αποφαίνεται για την περίπτωση υπερβολικού ελλείμματος. Νομίζω ότι αυτό είναι θέμα της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων. Όμως, θεωρώ ότι έχει δίκιο ο κ. όταν μας λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει μνήμα στον μηχανισμό χρηματοοικονομικής σταθερότητας. Διότι βεβαίως αυτά όλα έχουν επιπτώσεις όσον αφορά τον ετήσιο προπολογισμό και τις σχετικές οροφές τα οποία και μόλις συζητήσαμε στην Επιτροπή μας. Οπότε γι' αυτό θεωρώ ότι ε, το σημείο είναι δεν είναι δυνατόν να αποδεχθούν οι πολιτικές ομάδες παρά τη δυνατότητα τροπολογιών. Πάντως θεωρώ ότι Κατά τα άλλα, θα μπορούσαμε να εγκρίνουμε το κείμενο αυτό. Πάντω αν μπορείτε κύριε Πρόεδρε, δώστε μια παράταση μέχρι 17 του μηνό για τι τροπολογίες γιατί η προθεσμία που δίνεται τις 15 η του μηνό, εμεί θα πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει τι προτάσει μα για τον προβλημό του 2011 δώστε δύο μερούλε παραπάνω για να μπορέσουμε να ετοιμάσουμε τροπολογίες για αυτήν την έκθεση. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Θα σημειωθεί η πρότασή σας να μεταγενθεί η καταληκτική ημερομηνία από τις 15 στις 17 του μηνός. Εγώ δεν έχω καταρχήν αντίρρηση, αλλά προβλέπεται ψήφιση στην Επιτροπή των Υπολογισμών στην μαραθώνια σύνδεσή μας 27 με 29 Σεπτεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι οι τροπολογίες δεν θα έχουν μεταφραστεί, θα υπάρχουν μόνο σε μία γλώσσα. Δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί ότι θα γίνει σε όλες τις γλώσσες η μετάφραση. Ανδρέας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, ε, την έκθεση αυτή την έχουμε σε μία μόνο γλώσσα και τώρα έχει οριστεί η προθεσμία για τις 17. Ε, Νομίζω δεν υπάρχει πρόβλημα. Συμφωνώ με τον κύριο Γκαρίγκα. Και εγώ θεωρώ ότι όλο αυτό το θέμα των 60 δισεκατομμυρίων ευρώ, αυτό είναι το σημαντικό για μας στην Επιτροπή Υπεροπολογισμών ε, και από αυτού πρέπει να τοποθετηθούμε. Εκεί λοιπόν θα στραφεί και η προσοχή της δικής μου της ε, πολιτικής ομάδας. Ζητή άλλο το λόγο, κυρία ε, εισηγήτρια, θέλετε ξανά το λόγο. Ναι, πρόεδρε, ευχαριστώ. Δεν μπορώ να απαντήσω στον κύριο Φάρμ γιατί δεν μου είπε τι εννοεί, πού έχει ενστάσεις τώρα. Σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος ε, Γκαρίγα, Νομίζω ότι είναι σημαντικό, ακόμη και αν δεν είναι πρόκειτο περί αρμοδιότητος της δικής μας Επιτροπής, να ασχοληθούμε με τις ε, ε, ενστάσεις, να θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις επενδύσεις, τι γίνεται με όλα αυτά τα οποία μας ε, απασχολούν. Και άρα αν δεν προχωρήσουμε σε αυτή την πρόβληση των κυρώσεων δεν έχει νόημα. Ωραία, για τα 60 εκατομμύρια, αυτό που η κυρία Γένσεν, ε, χαίρομαι ότι θα ασχοληθεί. Ναι, όντω είναι θέμα σημασία υψίστη για τον προπολογισμό και αν η Επιτροπή Οικονομική έχει αναλάβει επί της ουσίας την αρμοδιότητα εμείς επίσης είμαστε συναρμόδιοι διότι στα πλαίσια του τοποθετικού προορισμού το 2007 το συζητήσαμε πριν από λίγο. ότι αν θέλετε να εξασφαλιστεί κάποιο είδου σταθερότητα στην ζώνη του ευρώ, θα πρέπει να, να, δούμε το κατά πόσον ε, θα αποφασίσαμε σε 9 Μαΐου, αν λειτουργούν, αν αποδίδουν όσον αφορά τους ε, επιχειρούντες τους, τους εμπλεκόμενους. Και αν δεν θέλουμε αυτό να είναι μόνο θέμα κρίση και θέλουμε να έχει πιο πάγιο χαρακτήρα, τότε αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να έχουμε κάποιο είδου ασφαλεί, σίγουρου ε, μηχανισμού από πλευρά ε, οικονομική και δημοσιονομική, διότι πιέζει η συγκυρία. Είναι τα πράγματα επίγοντα. Ε, έχουν λάβει κάποιε αποφάσει κυβερνήσει και έχουν δίκιο. Είναι θετικέ οι αποφάσει που Αλλιώ θα είχαμε μια καταστροφή. Πάντως, εδώ έχουμε κάτι που είναι εντελώς νέο. Και αν μέσω του προηγούμενου φροντίσουμε αυτά να εδραιωθούν, τότε θα έχουμε κάτι το πάρα πολύ χρήσιμο. Άρα, ε, σα προτείνω 17 Σεπτεμβρίου να είναι η καταληκτική ημερομηνία για τις προθεσμίες το μεσημέρι αυτή τη ημέρα για να προσπαθήσουμε έτσι να έχουμε ταυτόχρονα όσο γίνεται πιο πολλέ μεταφράσει για το κείμενο για τη συνέχεια. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια και πάμε στο σημείο 13 που είναι το τελευταίο που σήμερα θα συζητήσουμε διότι τα άλλα θέματα τα αναβάλαμε. Άρα έχουμε τον συνάδελφο και αντιπρόεδρο Κάλφιν που θα μας παρουσιάσει τα θέματα τα σχετικά με, τις, ε, με την εγγύηση στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Έχουμε τον κύριο Κρελιανκούρ, που είναι ο Διευθυντή για τι Διεθνεί ε, Υποθέσει τη Ευρωπαϊκή Τραπέζη ε, Επενδύσεων. Βρίσκεται εδώ, ναι, ναι, σηκώνει το χέρι ο κύριο Κρελιανκούρ. Καλώ ορίσατε και το λόγο πρώτα να λάβει ο κύριο Πρόεδρο. Κάλφιν. Συνάδελφοι, το θέμα αυτό αρχίσαμε να το συζητούμε γενικότερα. Σήμερα έχουμε ένα έγγραφο εργασία. Να κάτσουμε και να βρούμε λύση σε κάποια ζητήματα με εξωτερική ώρα τη σύνταξη του ελληνικού κειμένου. This proposal by the Commission, which is uh, very much based uh, on the wise persons group, which is uh, based on an external. Ξεκινούμε με κάποιες προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής από, επί τη βάση κάποιων ε, γνωμοδοτήσεων εξωτερικών συμβούλων και έτσι είπαμε ότι θα δούμε τι θα γίνει μέχρι το τέλος της παρούσης εντολής της ΕΤΕ του 2013. οι χώρες ΑΚΕ υπάρχουν σε άλλη συμφωνία, αλλά όλος ο βόλος κόσμος καλύπτεται από αυτή την εντολή. Η μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση προκύπτει από απόφαση του Συμβουλίου. Η σημερινή εντολή φτάνει μέχρι τον Οκτώβριο του 2011. Άρα, θα πρέπει χωρίς να έχουμε ένταση και στρες μια πλησιάζει αυτή η προθεσμία να προσπαθήσουμε να συμφωνήσουμε στα πλαίσια της συναπόφασης με το Συμβούλιο για την παράταση της εντολής μέχρι το 2013. Έτσι αυτές τις εξωτερικές δράσεις της ΕΤΕ θα πρέπει να υπόψη το οποίο προτείνεται στην έκθεση των σοφών. Υπό την προεδρία του Μισελ Καντεσί πρότειναν να υπάρχει ένα μεγαλύτερο, ευρύτερο πλαίσιο σε σχέση με το πώς η ΕΤΕ θα εξελιχθεί στο μέλλον. Πέραν του 2013, πολύ ενδιαφέρουσε μερικές προτάσεις σε σχέση με το τι πώς θα περιχαραγώσουμε το έργο της ΕΤΕ. Άρα να λάβουμε υπόψη κάποιες από τις προτινόμενες λύσεις και αλλαγές. Η πρόταση της Κομισιόν κατά τη γνώμη μου είναι μια πολύ καλή αφετηρία για να δουλέψουμε εδώ στο Κοινοβούλιο βάση είναι πάρα πολλές διαφορετικές γνώμες, όχι μόνο οι γνώμες της ομάδας των σοφών και των εξωτερικών συμβούλων, αλλά οι γνώμες και άλλων εμπλεκομένων, όπως τις χώρες, τις επιλέξιμες, μη παιδιά οργανώσεις, που όλοι αυτοί διαφέρονται πάρα πολύ όποτε συζητούνται τέτοια θέματα, όπως η εντολή της ΕΕΤ. Επίσης προτείνει εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πώς δηλαδή θα δημιουργήσουμε καλύτερες προϋποθέσεις συντονισμού μεταξύ της ΕΤΕ και των παραγόντων υλοποίησης των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αυτό είναι το, το οικονομικό όπλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να δούμε πόσοι πολιτικοί στόχοι της Ένωσης θα επιτευχθούν στα συγκεκριμένα μέρη του κόσμου. Γι' αυτό και έχουμε εδώ μια σειρά προτάσεων της Επιτροπής που είναι σημαντικές για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό το οποίο θέλουμε. Υλοποίηση των στόχων και κάλυψη της εντολής. Επίσης, έχουμε την πρόταση της Κομισιόν που μας οδηγεί σε πιο καλές προϋποθέσεις και όρους συντονισμού για τη λήψη αποφάσεων μεταξύ των διαφορετικών θεσμικών οργάνων από τη μία και της ΕΤΕ από την άλλη. Τρίτον, η πρόταση της Επιτροπής τώρα αποτελεί μια πιο λογική συνεκτική βάση για την εξωτερική αυτή δράση της ΕΤΕ, οριζόντιους υψηλού επίπεδου στόχου που θέτει και ταυτόχρονα κάποιε καθητήρες γραμμέ και πλαίσιο για τι διάφορε περιοχέ. Τώρα έχει επομένω μια καλύτερη πολιτική, πιο συνεκτική στον υπόλοιπο κόσμο από τη Ευρωπαϊκή Ένωση η Τράπεζα αυτή ήδη έχει αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε αυτές τις χώρες. θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε ότι μέχρι σήμερα ήδη έχουμε πετύχει. Με υπόψη τις προτάσεις της ΕΤΕ και εμείς που αξίζουν της προσοχής της ε, Επιτροπής μας για τις βασικές μας προτεραιότητες. Κάποια άλλα θέματα τα οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όταν έρθει η ώρα να αποφασίσουμε ή να ψηφίσουμε είναι το ότι πολλές φορές είναι συντηρητικές οι αποφάσεις του Συμβουλίου. Να μην τα πράγματα όσοι έχουν. Να λυθούν υπόψη κατά κάποιο τρόπο οι προτάσεις Κομισιόν, αλλά να μην θυγούν οι παλιές παράμετροι λειτουργίας της ΕΤΕ και άλλα δύο βασικά θέματα που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όταν έρθει η ώρα να αποφασίσουμε για την έκθεσή μας είναι πρώτον ο γενικότερος σκοπός της τράπεζας, της ΕΤΕ. Θέλουμε να της δώσουμε τη δυνατότητα να αποτελεί ταυτόχρονα και αναπτυξιακή τράπεζα. Αυτά προέρχονται και από την ομάδα Καμπτεσί και είχε πει μεσοπρόθεσμα ο κ. Καμπτεσί να δούμε πώς θα μπορέσουμε να συντονίσουμε τις διαφορετικές πολιτικές, τις διαφορετικές προσεγγίσεις στην ανάπτυξη. Αυτό είναι λοιπόν ένα από τα θέματα. Θέλουμε μια μεγαλύτερη δυνατότητα. Να μπορεί δηλαδή, γιατί να ασχοληθεί και με τους αναπτυξιακούς στόχους. Επίσης, το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να σκεφτεί και εναλλακτική λύση. Κάτι να υπάρξει εκτός ΕΤΕ. Ή να μην ασχοληθεί καθόλου σήμερα με αυτό το θέμα. Αλλά αυτό είναι το βασικά θέμα που θα πρέπει να συζητήσουμε. Δεύτερο θέμα είναι κάτι το οποίο αφορά τις οροφές. Που διέμπουν τη δράση της ΕΤΕ στις διάφορες περιοχές του κόσμου οι νέες χώρες, οι νέες επιλέξιμες χώρες θα έχουν ρύθμιση ίδιες οροφές όπως μέχρι τώρα. Επίσης, σε ορισμένε περιοχές έχει αναπτύξει δραστηριότητα μεγάλη η τράπεζα και ήδη έχουν καλυφθεί το 60% αυτών των οροφών πριν φτάσουμε σε αυτό το, στο μέσο της περίοδου της εντολής. Και μερικέ χώρε θεωρούν ότι έτσι θα είχε λιγότερε ευκαιρίε δράση η ΕΤΕ και μάλιστα σε κάποιε πάρα πολύ σημαντικέ περιοχέ του κόσμου, όπω α πούμε οι χώρε που γειτονιάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κάποια άλλα θέματα που θέλω να προσέξουμε. Ο θεσμικός ρόλος της ΕΤΕ σε σχέση με τις προτεραιότητες που θέτουμε. Ναι, γιατί να αυξηθούν οι αρμοδιότητες της Επιτροπής, αλλά θέλουμε οι αρμοδιότητες εξωτερικής δράσης να αυξηθούν. Γιατί κατά κάποιο τρόπο είναι ε, κάτι το οποίο μόλις τώρα το συγκροτήσαμε. Άρα, θέτοντας αυτούς τους στόχους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει την αρμοδιότητα της παρακολούθησης της απόδοσης και των αποτελεσμάτων της δράσης της ΕΤΕ σε χώρες εκτός Ένωσης. Επίσης, αν θέλουμε να έχουμε πιο ξεκάθαρους στόχους αναπτυξιακούς για την ΕΤΕ, θα πρέπει να έχουμε και πιο ξεκάθαρα κριτήρια για το πώς ορίζονται αυτοί οι στόχοι, να παρακολουθήσουμε την πορεία προς αυτούς τους στόχους, με ένα benchmarking. Εδώ, επομένως, ανακύπτουν πολλά θέματα. Άλλο θέμα. Συνεργασία με τα άλλα χρηματοοικονομικά ιδρύματα, την Παγκοσμία Τράπεζα ας πούμε, κάποιους αναπτυξιακούς εθνικούς φορείς, εμπορικούς ή μη, που ασχολούνται είτε με τραπεζικές υπηρεσίες είτε με την ανάπτυξη. Πολύ χρήσιμες οι προτάσεις γιατί λέει για κάποια πλατφόρμα που θα βοηθήσει για κάθε περιοχή να υπάρχει ένα συντονισμός σε σχέση με τη δράση σε συγκεκριμένη χώρα. Στο μέλλον θα το δούμε τις λεπτομέρειες, αλλά νομίζω θα πρέπει να αρχίσουμε να ασχολούμαστε με το θέμα, τουλάχιστον να βάλουμε το πλαίσιο της προβληματικής για αυτήν την πλατφόρμα. Γιατί ήδη υπάρχει πολύτιμη εμπειρία σε κάποιες περιοχές όπου ήδη έχει δράσει η ΕΤΕ και έχει συνεργαστεί με άλλα ιδρύματα. Κάτι άλλο που θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη είναι ο συνδυασμός των χορηγήσεων και δανείων πολλές φορές ο συνδυασμός αυτών δίνει περισσότερη προσβασιμότητα στα χρήματα της ε, ΕΤΕ. Και έτσι μπορεί να αναπτύξει μεγαλύτερη δράση η ΕΤΕ σε χώρες που δεν έχουν τρομερή επιστοληπτική αξιολόγηση. Έχουμε όμως πολύ την εμπειρία σε αυτό το τομέα. Και αν κανείς δει τις λεπτομέρειες, θα δει τα διμέρους θέματα που θα πρέπει να επιληθούν. Υπάρχουν τώρα κάποια άλλα θέματα όσον αφορά τη διαφάνεια, τη δυνατότητα μη κυβερνητικών οργανώσεων να υποπτεύουν τις δραστηριότητες των ε, αποδεκτών της, ε, των, των πόρων της ΕΤΕ, τα τελευταία χρόνια άλλωστε είχαμε μία βελτίωση όσον αφορά τον αποκλεισμό από τη συμμετοχή εταιριών που έχουν χρησιμοποιήσει φορολογικούς παραδείσους. Να, γιατί χρειάζεται η διαφάνεια και να πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε την πείρα της ΕΤΕ. Τέλος, ναι. Εντικά σας τα λέω ότι υπάρχουν πάρα πολλά σημεία. Απλώς λέω τα βασικά που θα πρέπει να συζητήσουμε. Είναι και το θέμα της παράτασης της εντολής. Έχουμε ένα αποθεματικό Δύο δις και έχει προταθεί αυτό να αποδεσμευθεί αυτό το κεφάλαιο και να πάει να καλύψει αυτή τη χορήγηση των εγγύσεων. Άρα να επιτρέψουμε στην ΕΤΕ να χρηματοδοτήσει προγράμματα και έργα για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος. Δεν είναι κακή ιδέα αυτό. Χωρίς να έχουμε συγκεκριμένα ανώρια Βέβαια να υπάρχει ισόρροπη αντιμετώπιση μεταξύ των διαφορετικών περιοχών και αν λοιπόν αποδεσμευτούν αυτά τα ποσά να δούμε εάν θέλουμε να έχουμε και επιπλέον προϋποθέσεις στις χώρες που θα διατεθούν αυτά τα χρήματα σε Ινδία, ας πούμε, σε Κίνα ούτως ώστε σε διάφορα φόρα οι χώρες αυτές να προσεγγίσουν τις θέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ή θα μπορούσαμε να αφήσουμε την εντεναδράση αυτές τις χώρες χωρίς να υπάρχει κανένας είδους τέτοια πολιτική δράση. Αυτά πρόεδρε είναι τα βασικά τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν. Πιέζει ο χρόνος σχετικά. Τα λέει το κομπουνιούς όλα. και να προσπαθήσουμε να σας διαβιβάσουμε την έκθεση τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου και πριν να ολοκληρώσουν το έργο τους οι πολλές συναρμόδιες επιτροπές του Κοινοβουλίου. Κάνω ό,τι μπορώ να συντονιστώ με τους συναδέλφους της άλλες επιτροπές. Και προσπαθώ να κάνω τις επαφές με τους άλλους εμπλεκόμενους και όταν έρθει η ώρα να έχουν κλείσει όλα αυτά τα οποία σας είπα ότι κρεμούν. Και να έχουμε καταλήξει κάποια λύση αποδεκτή. Και αν τελικά συμφωνήσουμε το Συμβούλιο, θα πάμε σε ψηφοφορία στην Σύνοδο του Ιανουαρίου. Και αν πάμε σε συνδιαλλαγή, αυτό θα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε πάλι τον Ιανουάριο για να έχουμε ολοκληρώσει το αργότερο τη διαδρομή μας την άνοιξη του χρόνου. Αλλιώς θα έχει πρόβλημα να δουλέψει η ΕΤΕ εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά έχουν να πω Να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προχωρήσει το θέμα όσο γίνεται καλύτερα γιατί είναι πολύ σημαντικό. Très bien, merci monsieur le δεν έχει ζητήσει κανεί το λόγο. Α, όχι, η Έλγα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ε, κάνατε όλη αυτή την ομιλία και μας δώσατε και τις ε, πληροφορίες. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για το ποια θα είναι η μολυντική πολιτική επενδύσεων ε, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ποιο είναι το πεδίο, κατά πόσον θα πρέπει να υπάρξει συνεχρηματοδότηση ή όχι. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα Υπάρχει η πολιτική διαμάχη, αν θέλετε, ανάμεσα στη Γαλλία και τη Γερμανία για το κατά πόσον ε, θα πρέπει να υπάρχουν ρυθμίσεις, πολιτικές ρυθμίσεις για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή όχι. Και ρωτώ, εσείς αυτό το θέμα ε, το θίγετε στην εκθεσία ή μήπως η εκθεσία δεν ασχολείται ε, με αυτό το θέμα. Μιλάμε για την ΕΤΕ, όχι για την Κεντρική Τράπεζα. Υπάρχει μια μικρή διαφορά. Um, Δεν ζητά κανείς άλλο στο λόγο. Εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Και όπως και εκείνος να υπογραμμίσω την πολιτική σημασία του διακυβεύματος. Όπως μας θύμισε, η ομάδα των σοφών, της οποίας προείδρευε ο πρώην Γενικός Διευθυντής ε, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, κ. Γιανσού, είχε την ευγένεια να έρθει εδώ στην Επιτροπή Προπολογισμών για να μας παρουσιάσει τα πορίσματά του πριν να τα δημοσιεύσει και πριν και να τα επιδώσει στην Κομισιόν, η οποία στη συνέχεια επεξεργάστηκε το σχέδιο κανονισμού. Και υπάρχουν πολλές ε, πολιτικά ενδιαφέρουσες πτυχές Ιδιότερα σε μια περίοδο που όπως έδειξαν τα υποψηνές συζητήσεις, το χρήμα σπανίζει και κοστίζει. Όλα είναι και περισσότερο. Άρα λοιπόν δεν θα με εντυπωσίαζε τα τρία θεσμικά όργανα είτε να συμφωνήσουν στην ε, συνδιαλλαγή είτε να πρέπει περισσότερο να προωθηθεί η ΕΤΕ για να χρηματοδοτήσει κοινοτικά προγράμματα. Ε, άρα λοιπόν φυσικά δεν είναι αντίθετο να πούμε στον κανονισμό πώς θα κατανεπιθούν ανάμεσα στα εσωτερικά και εξωτερικά σχέδια τα χρήματα της ΕΤΕ, αλλά αυτό είναι μια βάση, είναι μια πλατφόρμα για τη δική μας συζήτηση για το μέλλον της ΕΤΕ και των δράσεών της εκτός της Ένωσης. Αυτά θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας. Και έπειτα, όπως είπε και ο κύριος Καλφίν, η βοήθεια προς προγράμματα σε αναπτυσσόμενες χώρες ήδη είναι ρόλος πολλών ε, χρηματοδοτικών οργάνων, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, οι περιφερειακές, οι περιφερειακές και θεσμοί που υπάρχουν σε όλες τις υπήρους και θεσμούς που, είναι, που προγραμματίζονται τον Νοέμβριο. Προβλέπεται, αν όλα πάνε καλά από πολιτικής άποψης, μια νέα διάσκεψη κορυφής της Ένωσης για την Μεσόγειο και ένα από τα θέματα που είναι επιτάπητος είναι η δημιουργία μιας τράπεζας για την Μεσόγειο. Τώρα θα ληφθεί απόφαση ή όχι, Θα έχει σχέση αυτό το νέο μέσο, το νέο εργαλείο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή όχι. Θα πρέπει δηλαδή να σκεφτούμε και να χρησιμοποιήσουμε τα κατάλληλα εργαλεία πριν να δημιουργήσουμε νέα. Και, εν πάση περιπτώσει, να σκεφτούμε τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι νέες δυνατότητε που δίνονται στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στο πλαίσιο αυτού του κανονισμού θα λειτουργήσουν σε αρμονία με τα όσα ήδη υπάρχουν με άλλα ή από άλλα θεσμικά όργανα που θα δημιουργηθούν. Υπάρχει επίσης το θέμα, όπως είπε και ο κύριος Καλφίν, το θέμα των όρων, των πολιτικών όρων για τα δάνεια. Πολύ λεπτό ζήτημα. Επί το οποίο μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν ποτέ πολύ αποτελεσματική όσον αφορά δηλαδή τα χρήματα που δίνει στην αναπτυξιακή βοήθεια που χρηματοδοτείται από, τις, από τον κοινωτικό προπολογισμό. Έχουμε υπογράψει διάφορα άρθρα που υποτίθεται σκληραίνουν τους όρους, ε, αλλά στην πράξη κυρώσεις πολύ σπάνια έχουμε ε, επιβάλει. Όταν πρόκειται για δάνεια όμως ο πολιτική άποψη είναι διαφορετικό γιατί ένα δάνειο δεν είναι πραγματικά ενίσχυση, δεν είναι βοήθεια. Είναι θεμητό όταν δίνουμε ένα δάνειο να θέτουμε και κάποιον πολιτικό όρο. Επισήμως όχι. Αν επισήμως θα πρέπει να δούμε. Και φυσικά για ένα τέτοιο θέμα οι θύνοντες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων θα έχουν και αυτή λόγο. Γιατί υπάρχει και μια κάποια διοντολογία που διέπει τις πρακτικές της Παγκόσμιας Τράπεζας αλλά και άλλου οργανισμού τέτοιου τύπου, καθώς και για την Ευρωπαϊκή ε, Τράπεζα Επενδύσεων και δεν μπορούμε να μην το λάβουμε υπόψη. Αναφέρω λοιπόν όλα αυτά τα ζητήματα, απλώς και μόνο για να υπογραμμίσω τη σημασία των όσων είπε ο εισηγητής μας. Και να σας πω ότι αφού έρχεται αυτή τη στιγμή, αυτή η πρόταση έχει ιδιαίτερη ε, σημασία. Λοιπόν, δεν ζητά κανεί το λόγο να πούμε λοιπόν ότι αυτή η θέση του εισηγητή μα είναι αποδεκτή. Κύριε Διευθυντά, θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο. Ναι, ευχαρίστω κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι αυτά τα οποία μόλις τώρα είπατε και αυτά που είπε και ο εισηγητής είναι βεβαίως πάρα πολύ σημαντικά για μας και θέλω να επενθυμίσω στην Επιτροπή ε, τι ακριβώς κάνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, εμείς ε, εφαρμόζουμε τις εντολές που μας έχει δώσει ε, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Άρα, δηλαδή, στηρίζουμε τον πολιτικό προσανατολισμό. Και αυτό ίσως είναι απάντηση στο ερώτημα που θέσατε στην αρχή σχετικά με τους όρους. Γιατί, πράγματι, και την επιλεξιμότητα. Δεν είναι το ίδιο να πει κανείς, όταν αποφασίζει κανείς για χορηγήσεις ή για δάνεια, όταν πρόκειται για την κλιματική αλλαγή, για την βελτίωση της απασχόλησης, για την αλλαγή του ρου της μετανάστευσης. Αυτή είναι στόχη της Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή η όροι, αυτοί είναι και η όροι για να δοθούν οι χορηγήσεις. Πράγματι, οι εγγυήσει που δίδονται από τον προπολογισμό, αυτό είναι κάτι που δεν έχει στοιχήσει ούτε ένα ευρώ στον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Την ίδια στιγμή όμως για την τράπεζα ε, έχει καταστεί αφές να ε, με αυτές τις εγγύησεις. Αυτό λοιπόν λειτουργεί πάρα πολύ καλά και γι' αυτό εμείς ε, προτιθέμεθα να χορηγούμε αυτά τα δάνεια από κοινού με την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Ε, κύριε Σιγητά, όσον αφορά την ουσία των θεμάτων, εμείς εξετάζουμε, εμείς χαιρόμεθα που εξετάζετε αυτά τα θέματα που και εμείς θεωρούμε πολύ σημαντικά. Ε, δεν θέλω τώρα ε, να δαπανίσω χρόνο για να αφαιρθώ σε όλα αυτά. Θέλω μόνο να πω ότι το θέμα της ανάπτυξης είναι πολύ σημαντικό. Και επαναλαμβάνω αυτά που είπε ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ε, στην έκθεσή του. Δηλαδή, αν μας ζητήσουν να πράξουμε αν μας ζητηθεί να πράξουμε περισσότερα στον τομέα της ανάπτυξης, παρακαλώ δώστε μας και τους πόρους. Και πόρους δεν είναι μόνο το ανθρώπινο δρομικό, είναι και πρόσβαση ε, στις πιστώσεις. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς ε, δάνεια. Ε, θέλω λοιπόν να υπογραμμίσω ότι η λέξη αποτελεσματικότητα που εμφανίζεται αρκετές φορές στο σχέδιο της έκθεσης κατά την άποψή μας ίσως να μην είναι και η καλύτερη. Γιατί εμείς πιστεύουμε μπορούμε να αποδείξουμε ότι είμαστε τόσο αποτελεσματικοί που μερικές φορές ε, αυτό δημιουργεί προβλήματα κυρίως όταν δεν υπάρχουν οι πόροι. Τώρα, όσον αφορά τα ανώτατα όρια, θέλω να πω ότι η ΕΤΕ εκατέβαλε μία προσπάθεια να ανταποκριθεί ε, στην κρίση κατά τα τελευταία δύο χρόνια και με τον τρόπο αυτό ίσως ε, να προέκυψε ε, ένα χάσμα σε σχέση με τα ποσά που εκταμιεύτηκαν σε τελική ανάλυση. Όσον αφορά το ρόλο του Κοινοβουλίου, Πράγματι, εμείς ε, θεωρούμε ότι είναι σωστό και να οριστούν οι στόχοι και να γίνεται και αξιολόγηση των επιπτώσεων. Ίσως ε, έχουμε κάποια δυσκολία στην πρακτική. Αν το Κοινοβούλιο επιθυμεί κάποια διατύπωση να συμπεριληφθεί και στην εκτέλεση του σχεδίου, γιατί αυτό καλύτερα να το κάνουμε εμείς και εσείς μετά να μας κρίνετε κατά πόσον έχουμε επιτύχει τους στόχους μας. η συνεργασία με τους διεθνείς οργανισμούς. Ε, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για μας. Και όσον αφορά τη διαφάνεια και την αντιμετώπιση των ε, εξωχώριων ε, χρηματοπιστωτικών κέντρων, νομίζω ότι γνωρίζετε ότι η ΕΤΕ προηγείται, παίζει πρωτοπόρο ρόλο σε αυτόν τον τομέα. Και μερικές φορές αυτό οδηγεί σε δυσκολίες όταν προβαίνουμε σε συγχρηματοδότηση με άλλους. Γιατί αν εμείς δεν μπορούμε να επιβάλλουμε όλους τους όρους, ε, τότε και οι υποφελούμενες ε, χώρες έχουν περιθώριο λιγμών. Αυτό δεν είναι καλό. Όσο πιο γρήγορα ε, ταυτιστούμε όλοι σε μία γραμμή, τόσο καλύτερα. Πράγματι, όσον αφορά την Κοπενχάγη, αυτό είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και με την έκθεση, αλλά θα ήθελα να σε επισημάνω ότι όταν παραδείγματο χάρη ε, δραστηριοποιηθήκαμε στην Κίνα, αυτό δεν έγινε επειδή οι Κινέζοι χρειαζόντουσαν χρήματα, αλλά διότι εκτιμούν δύο πράγματα που μπορούμε να προσφέρουμε. Το ένα είναι η τεχνογνωσία και αυτό ε, μας το είπαν. Ε, μας λένε ότι εσείς μπορείτε να μας βοηθήσετε να επιλέξουμε τα προγράμματα που είναι σημαντικά και όχι οτιδήποτε. Έτσι λοιπόν ε, προσφέρουμε υποστήριξη με τη μορφή της ε, τεχνικής ανάλυσης και μην ξεχνάτε, εμείς έχουμε και τη δική μας την τεχνολογία. Άρα λοιπόν και αυτά θα πρέπει να ε, λάβετε υπόψη όταν θα κάνετε την τελική αξιολόγηση. Αυτά. Η Κομισιόν δεν επιθυμεί να λάβει το λόγο. Κύριε Σιγητά, εσείς θέλετε να ξάγετε τα συμπεράσματα. Νομίζω πως θα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στο μέλλον. Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με τα όσα είπε ο κύριος Διευθυντής αφορά την αποτελεσματικότητα των κοινοτικών πολιτικών και το ρόλο της τράπεζας στην εφαρμογή των πολιτικών αυτών. Εδώ βεβαίως και δεν αναφερόμουν στην αποτελεσματικότητα της, ε, του οργανισμού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και γι' αυτό και όταν μιλάμε για το ρόλο του Κοινοβουλίου ακριβώς αυτό πρόκειται για τον ορισμό, καθορισμό πολιτικών και την εξέταση των αποτελεσμάτων για το πώς δηλαδή η ΕΤΕ συνέβαλε στην επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων. Συμφωνώ Συμφωνώ λοιπόν απόλυτα με τα όσα μόλις είπατε. Και νομίζω πως ε, θα έχουμε επικοδομητικές ειδήσει και στο μέλλον. Ευχαριστούμε κύριε Σιγητά. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, Κύριε Σιγητά, η πρότασή σας αντιστοιχεί στα όσα έχουμε βάλει στο κομπούνιος. Δηλαδή, υποβολή σχεδίου εκθέσεως 27 Οκτωβρίου, γιατί μέχρι τότε θα ε, ασχοληθούμε από τον προπολογισμό 2011. Ε, υποβολή ε, των τροπολογιών 4 Νοεμβρίου, 4 Νοεμβρίου και ελπίζουμε ότι θα υιοθετηθεί την 1η Δεκεμβρίου γιατί ε, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι τρεις επιτροπές που θα γνωμοδοτήσουν θα πρέπει να δώσουν τις νομοδοτήσεις 25 με 26 Οκτωβρίου. Υπάρχουν και άλλες δυο στις οποίες θα ζητήσουμε να γνωμοδοτήσουν στις ίδιες προθεσμίες. Αν δεν ζητά κανεί άλλο το λόγο, νομίζω πω ε, ολοκληρώσαμε την εξέταση τη ημερήσια διάταξη. Είδατε τα έγγραφα που έχουν διανεμηθεί ενημερωτικά και σα θυμίζω ότι η επόμενη μα συνεδρίαση ορίζεται, είναι η μαραθώνια συνεδρίαση 28-29-30 Σεπτεμβρίου και είναι πιθανό, θα το αποφασίσουμε απόψε οι συντονιστές, να κάνουμε και μια επιπλέον συνεδρίαση τη Δευτέρα το βράδυ, την επόμενη Δευτέρα, στο Στρασβούργο. Την πρώτη μέρα της Ολομέλειας. Θα το αποφασίσουμε απόψε το βράδυ. Θα το ξέρετε αύριο το πρωί. Κύριος Άγκλουντ, στα διάφορα. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Μια πρακτική ερώτηση. Είναι δυνατόν να καταθέσουμε ε, τροπολογίες για την κινητοποίηση του, Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, δεδομένου ότι αναβλήθηκε η εξέταση της έκθεσης αυτής της κυρία Ματέρα. Μπορούμε να καταθέσουμε τροπολογίες. Όχι, δεν, έχουμε, δεν υπάρχει προθεσμία. Θα σας το... Θα σας διαβιβάσουμε μόλις θα έχουμε ορίσει προθεσμία. Ευχαριστώ πολύ. Τέλος συνεδρίασης. Θα μείνουν μόνο οι συντονιστές. Διακόπτουμε για λίγο λεπτά οι συντονιστές να μείνουν στην αίθουσα για να εκμεταλλευτούμε για ένα τεταρτάκι του διερμηνείς.